όπου θα πρέπει να προσθέσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας Αλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές είναι ο μόνος δωρητής εκτός από τα τέσσερα κράτη στα οποία ανήκουν τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα. Επίσης, τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα είναι επιλέξιμα για τα οριζόντια μας προγράμματα που αφορούν όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Τα προγράμματα αυτά είναι ανοιχτά για τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα, εκτός από τις ειδικέ διατάξεις που διέπουν ορισμένα προγράμματα. Καταρχήν όμως είναι επιλέξιμα αυτά τα υπροπόντια εδάφη και διαμερίσματα, όπως μέσα στα πλαίσια της έρευνας και της καινοτομίας. Υπάρχουν όμως και γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το περιβάλλον και την βιοπικιλότητα, όπου τα υπερπόντια διαμερίσματα έχουν πρόσβαση, αλλά με εκδήλωση ενδιαφέροντος και με υποβολή προγράμματος. Μπορούν λοιπόν να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Ένας άλλος τρίτος τρόπος συμμετοχής και οι επόμενοι ομιλητέ θα το αναπτύξουν αυτό το θέμα, αφορά τις εμπορικές σχέσεις, το εμπορικό τμήμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στα διαμερίσματα ένα ειδικό εμπορικό καθεστώς το οποίο είναι πολύ πιο ε, πλεονεκτικό και ευεργετικό σε σχέση με τους άλλους εταίρους. Ο κύριος Ράμκοβαλ θα σας μιλήσει για τις ε, γενικές κατευθυντήριες γραμμές και την εμπορική πλαισίωση που διέπει τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε τα υπερπόντια εδάφη με ένα πολύ πλεονεκτικό καθεστώς. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει υποβάλει μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που είναι απότοκη μίας μακροχρόνιας διαδικασίας. Άρχισε το 2008 με την πράσινη βίβλο, όπου, οπότε και άνοιξαν οι διαβουλεύσεις. Το 2009 είχαμε μία ανακοίνωση της ε, Κομισιόν για τις προτεραιότητες μέχρι το 2013 και πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο απετέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων μέσα στα πλαίσια του φόρουμ ε, υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, με εκπροσώπους από τα υπερπόντια εδάφη και εκπροσώπους από τα κράτη-μέλη. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε και άλλες εκδηλώσεις υπέρ των υπερποντίων εδαφών και διαμερισμάτων το 2011 τα υπερπόντια εδάφη υποστήριξαν ένα κοινό κείμενο με τα τέσσερα κράτη-μέλη, τονίζοντας την άποψη και τις φιλοδοξίες αυτής της σύνδεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δική της πλευρά διενέργησε αρκετές μελέτες, είτε εσωτερικές είτε με εξωτερική ανάθεση, που ε, τόνωσαν τις εργασίες ως προς την ανάλυση αντικτύπων, ανάλυση αντικτύπου μέχρι τον ε, Μάρτιο-Απρίλιο του 2012. Πρόκειται για μελέτη αντικτύπων που βοήθησε την Επιτροπή να συντάξει την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου σε στέρες βάσεις. Σήμερα, το Σεπτέμβριο 2012, προβλέπεται το φόρουμ, ε, σε μια εβδομάδα δηλαδή θα γίνει αυτό το φόρουμ υπερπόντιων διαμερισμάτων και Γρυλανδίας, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και τα 26 υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα θα μπορέσουν να λάβουν θέση. Στη συνέχεια αυτού του φόρουμ θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μέσα στα πλαίσια των χωρών και του Συμβουλίου, που θα δώσουν συνέχεια σε αυτή την πρώτη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για μία παρουσίαση σε γενικές γραμμές μόνο. Η πρόταση βασίζεται σε τρεις αρχές. Πρώτη αρχή. Ο μύτος της Αριάδνης αφορά την, τον εξυγχρονισμό, τα κοινά συμφέροντα και τη συγκέντρωση σε εκείνα προγράμματα. Η Επιτροπή κατά τα τελευταία φόρα ανάπτυξε αυτά, αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι έγινε από το 2001 και μετά. Από τότε που η Συμφωνία Σύνδεσης τέθηκε σε ισχύ ως προς το εμπορικό της σκέλος και την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσης, θέλουμε να υπάρχει σωστότερη χρηματοδότηση και κοινοτική μόχλευση, προβάλλοντας μία ε, συγκέντρωση θεμάτων και συγκέντρωση πόρων, τονίζοντας κοινά συμφέροντα που αφορούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπερπόντια διαμερίσματα. Μιλάμε για μια κοινή θεματική λοιπόν, η οποία δεν απέχει από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η βιοπικιλότητα, το περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν παρά ένα μόνο παράδειγμα, το οποίο καταδεικνύει τι εννοούμε όταν μιλάμε για κοινά συμφέροντα. Η διάρθρωση του κειμένου της Επιτροπής, της πρότασης της Επιτροπής έχει αλλάξει σε σχέση με τα κείμενα που είχαμε μέχρι τώρα. Περιλαμβάνει πέντε τμήματα, αποτελείται από πέντε τμήματα. Καταρχήν οι γενικοί κανόνες, οι γενικές ρήτρες και διατάξεις, δεύτερο τμήμα. Αφορά τους τομείς συνεργασίας, όπου ασχολούμεθα με το βιοεμπόριο ή τους ε, άλλους τομείς παραγωγής. Εδώ θέλαμε να ομαδοποιήσουμε τους διάφορους τομείς ε, δυνάμεις συνεργασίας. Το τρίτο τμήμα που αφορά αποκλειστικά το εμπόριο και τα συναφή ζητήματα. Το τέταρτο τμήμα που μιλά για τα μέσα και μηχανισμούς που θα κινητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη αυτών των εδαφών και ένα τελευταίο τμήμα που αφορά τις ρήτρε μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας Σύνδεσης και τι μπορεί να γίνει όταν αλλάξει το καθεστώς ενός υπερπόντιου εδάφους και αν αυτονομηθεί. Υπάρχουν και τα παραρτήματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την απόφαση, δεν είναι προσαρτήματα της απόφασης Πρόκειται για τους κανόνες θέση εφαρμογή του εμπορικού σκέλους. Θα σταματήσω εδώ. Σας έκανα μια γενική εισήγηση αυτής της πρότασης και νομίζω ότι στη συνέχεια θα μπούμε σε λεπτομέρειες ως προς τα τμήματα αυτής της πρότασης νομοθετικού περιεχομένου και με μεγάλη χαρά θα απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ήξερα λίγο τις ε, προτάσεις Κομισιόν, αλλά ε, δεν τις είχαμε συζητήσει ως τώρα. Θα γίνει αυτή η συζήτηση κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Ο λόγος στην κυρία Κλοέ Καλβινιά πρόεδρο της Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωση Υπερπόντιων Χωρών και ε, Εδαφών. Κυρίε και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης για την διοργάνωση αυτής της ακρόασης, και για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μωρίς Πονγκά επίσης, Ευρωβουλευτή, για την συνεχή εργασία του να φέρει τα θέματα των ΙΧΕ, των υπερπών χωρών και έδαφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης όλους τους συνδιοργανωτές του. Μετά τον κύριο Σαραμόντη, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ ω ε, ε, πρόεδρο τη ΟΚΤΑ, τη Ένωση δηλαδή ε, όλων των υπερπόνιων χωρών και εδαφών που ανήκουν στην Γαλλία, θα ήθελα να σας δώσω εγώ την ε, δική μας, το δικό μας όραμα για την σύνδεση αυτών των χωρών και των εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επαναλάβω ε, ορισμένα ελάχιστα στοιχεία που είπε ο κ. Σαραμόντη, συζητώ συγγνώμη. Ε. Σίγουρα έχουν πολλά κοινά σημεία και πολλές διαφορές οι, οι χέοι, τα υπερπόντες χώρες και εδάφη. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως από μια διαπίστωση απλή ότι η οικογένεια των είχε ε, είναι σχετικά άγνωστη στις Βρυξέλλες. Είναι μια οικογένεια που ταλαιπωρείται από την έλλειψη ορατότητας. Είναι οι Ευρωπαίοι γείτονες των άκρο ε, άκρος περιφερειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι χώρες ΑΚΕ και χώρες μία ΑΚΕ δεν είναι τρίτες χώρες, ε, δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι χώρες και εδάφη συνδεδεμένα. Δεν, γνωρίζονται, δεν τις γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά στις Βρυξέλλες. Η θέση τους είναι πολύ δύσκολη. Στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ε, υπάρχει μια μονάδα που ασχολείται με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ασχολείται με, και με τις ΙΧΕ. Στο Συμβούλιο η Επιτροπή ΑΚΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή ΔΕΒΕ. Οι ΙΧΕ δεν έχουν τους ίδιους στόχους με τις αναπτυσσόμενες χώρες όμως. Παρόλο ότι στην ισχύουσα συμφωνία σύνδεσης ε, γίνεται λόγος για τις λιγότερο ανεπτυγμένες ΙΧΕ. Πλην όμως δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι ο εξή. Οι ΙΧΕ δικαιούνται της χρήσης του ίδιου χρηματοοικονομικού μέσου με τι ε, ε ΑΚΕ, αλλά το, δηλαδή το ΦΕΔ, το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, όμω είναι αρκετό αυτό. Ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά την περίοδο μετά το 2013 είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση. γνωρίζουμε ότι είναι ε, ευρωπαϊζουσε ε, χώρες και εδάφη, ε, είναι βιτρίνα της Ευρώπης, ανήκουν σε δύο κόσμου, είναι ακόμα πιο απομακρυσμένες και από τις άκρως περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι κοινά χαρακτηριστικά τους και, και τα συνδέουν αυτά τα έδαφη και αυτέ τι χώρε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, είναι μια οικογένεια την οποία δεν γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά είναι και πολυπληθής οικογένεια. Το είπε ο κ. Σαραμόντης. Χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία, το είπαμε και αυτό, διαφορές στον πληθυσμό, στην έκταση, στον βαθμό αυτονομίας τους σε σχέση με τις χώρες με τις οποίες είναι συνδεδεμένες και βέβαια διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Μεγάλη ποικιλία Βασικός τομέα, βασική τομή τομή είναι οι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε, οι ε, υδατοκαλλιέργειε, ε, η εκμετάλλευση φυσικών πόρων, η αλληλεία και ο τουρισμό. Υπάρχουν όμως και κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Ε, όλοι οι κατοικοί του κατά κανόνα είναι, έχουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. όλα είναι νησιά. δεν είναι χώρες έχουν τις περισσότερες φορές στρατηγική θέση και είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Από πλευρά περιβάλλοντος, οικονομίας έχουν σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και όλες οι χώρες και τα διαμέσματα αυτά είναι ευκαιρίες, αποτελούν ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση είχε ε, θα κλείσει 10 χρόνια του χρόνου και έχει ως ε, στόχο να προσπίσει τα συλλογικά του συμφέροντα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εργάζεται με βάση μια προεδρία η οποία αλλάζει κάθε χρόνο. Φέτος είναι πρόεδρος, ο πρόεδρος της Γρυλανδίας, ο κ. Κλάιστ. Υπάρχει και το φόρουμ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΧΕ. τέσσερα κράτη-μέλη, εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ευρωβουλευτέ ε, και αντιπρόσωποι τη Προεδρία κάθε φορά. Στο φετινό φόρουμ θα είναι η Προεδρία τη Κύπρου. Ε, από το τέλο του χρόνου, ο πρόεδρο του Σαν Πιέρ και Μικλόν θα γίνει πρόεδρο τη Ένωση. Η ΟΚΤΑ, η Ένωση ΧΕ, θα αποκτήσει αντιπροσωπεία στι Βρυξέλλε πολύ σύντομα το γραφείο στις Βρυξέλλες ε, υπάρχει ήδη βέβαια από το 2006 αλλά θα κινητοποιηθεί πολύ περισσότερο στο μέλλον. Επόμενο σημείο στο, το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι το ενδιαφέρον των ΙΧΕ για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία τη θέλουν να την προωθήσουν. Οι ΙΧΕ έχουν ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς πολύ ισχυρούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, υπογραμμίστηκε από το 2008 στην ανάλυση που είχε γίνει, ένα μεγάλο αριθμό από τις ηχεία εφαρμόζουν de facto το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ορισμένες συχέ όπως το Σέμπιαρ και Μικλό ε, χρησιμοποιούν μάλιστα και το ευρώ. Η οικονομική και τεχνική υποστήριξη τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, ε, αναπτυξιακή της πολιτική έχει σημαντικές θετικές συνέπειες. Αυτό αποδείχθηκε σε μια έκθεση, σε μια ανάλυση που έγινε από το 2009 στο 2009. η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σημαντική προστιθέμενη αξία να δώσει και δίδει ήδη με την ενίσχυσή της. Η, έχουν συμμετάσχει στην ανάλυση που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια με την πράσινη βίβλο. Ε, μετά συμμετείχαμε ε, στις διάφορες αξιολογίες που έγιναν, πολιτικά ψηφίσματα ετήσια από πλευράς ε, Ένωσης είχε και από το 2011 ακόμα πιο ενεργά. Απόδειξη αυτού του ενδιαφέροντος είναι ότι πολυάριθμες είχε ε, διαφημίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Καλυδονία, για παράδειγμα, διοργανώνει μια ε, ε, εβδομάδα κινηματογράφου, πολιτιστική εβδομάδα. Έχουμε το, στην Αρούμπα το σπίτι της Ευρώπης και πολλές άλλες πρωτοβουλίες η Ευρώπη δεν ακούγεται και πολύ εκεί πέρα, οπότε είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δρασει. Υπάρχει ένα γραφείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουμαία, που καλύπτει τέσσερι χώρες και εδάφη τη περιοχής και από ό,τι φαίνεται η Κομισιόν σκέφτεται να το κλείσει και όλα αυτό μας ανισχύει ιδιαίτερα. Ε, θα ήθελα επίσης να σας δώσω τρία παραδείγματα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εξαιτία ε, της έλλειψης αναγνώρισης του ευρωπαϊκού μας χαρακτήρα και, της, ε, και το, του ευάλωτου χαρακτήρα μας. Ε, είχαμε πετύχει γενική ε, πρόσβαση σε όλα τα οριζόντια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς ε, για να τονιστεί αυτή η, ο σύνδεσμος ανάμεσα στη, στη ΣΥΧΕ και στα Ευρωπαϊκή Ένωση όμω, αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερα προβλήματα στην, στην πράξη, στην πρόσβασή μας. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα LIFE, στο οποίο δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε πρόσβαση μέχρι τώρα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ο πολιτικός στρατηγικός διάλογος. Ε, είχε με την υποστήριξη των κρατών μελών έχουν ανάγκη να παρακολουθούν από κοντά ε, την αναθεώρηση της ε, περιφερειακής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για παράδειγμα με, τις, με, τον, ε, με τις χώρες του Ελληνικού Ωκεανού, με τις χώρες της Καρεβικής ε, κλπ. για να προσαρμοστεί στις ε, κλιματικές αλλαγές. Ε, πρέπει επίσης να μπορούν να παρακολουθήσουν το διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα όργανα ολοκλήρωσης της κάθε περιοχής και να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη τους στις διαπραγματεύσεις και στις δράσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ο, ο προγραμματισμός βοήθειας. Η, αυτή τη στιγμή ε, χαίρουν κάποιων απλοποίησεων, οι οποίε όμω δεν είναι αρκετέ σε ό,τι αφορά την χρηματοδότησή του. Ζητούν εδώ και αρκετό καιρό ε, ένα προτιμησιακό καθεστώ σε αυτό το θέμα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανάπτυξης ε, που έχει ως βασικό στόχο της χώρας ΑΚΕ ε, και κυρίως για την καταβολή της φτώχεια. να αναφέρω μόνο ότι στην κοινή θέση του 2011 τα κράτη-μέλη και είχε είχαν ζητήσει να δημιουργηθεί ένα ειδικό μέσο, χρηματοδοτικό μέσο, που ε, θα έχει ως ελάχιστο στόχο την απλοποίηση και την προσαρμογή ε, των διαδικασιών που αφορούν τη ΣΥΧΕ. Σήμερα, οι διαδικασίες προγραμματισμού μπορούν να διαρκέσουν και τρία και τέσσερα χρόνια. Θα τελειώσω αυτή μου την εισαγωγή με μια γενική τοποθέτηση για την νομοθετική πρόταση ε, σε σχέση με τα αιτήματα που ε, είχαμε εκφράσει το 2011. Χάρηκα που άκουσα ότι η Επιτροπή ε, Ανάπτυξης θα ετοιμάσει μια έκθεση για το θέμα αυτό. Η πολιτικό ψήφισμα θα υιοθετηθεί στην υπουργική διάσκεψη 25 Σεπτεμβρίου από τις ΙΧΕ. Θα τονιστεί ιδιαίτερα το θέμα της πράσινης ανάπτυξης, η εκπαίδευση, η καινοτομία και η έρευνα. Ε, σε αυτού του τομεί η πράσινη ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη των ΙΧΕ. Όμω σε αυτά τα συμπεράσματα θα συμπεριλάβουμε και πολιτικά μηνύματα για την νομοθετική πρόταση για τι ΙΧΕ, την οποία πήραμε μέλο Ιουλίου. Ε, δεν μπορώ να σα πω ακριβώ ποια θα είναι τα συμπεράσματα αυτά, αλλά να σα πω τι περίπου θα περιλαμβάνουν. Καταρχήν, ε, θα εκφράσουμε μια γενική ικανοποίηση από πλευρά των ΙΧΕ για αυτή την πρόταση που έλαβε υπόψη πράγματι την ανάγκη αναθεώρηση του στόχου τη εταιρική σχέση να σας υπενθυμίσω ότι η θέση μας έλεγε πως ε, χρειάζεται μια συνεχής οικονομική ενίσχυση ε, λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς ε, στόχους και την, ε, το ευάλωτο ε, της, ε, τον είχε. Ευχαριστούμε πολύ την Κομισιόν για αυτή τη δουλειά που έκανε για την αναθεώρηση της απόφασης. Είχε, επίσης θα ε, εντοπίσουν συγκεκριμένα σημεία της ε, πρότασης τα οποία θα ήθελα να τονίσουν. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, η, τα, πρέπει να ενισχυθούν τα όργανα της Ένωσης και να διοργανωθούν στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης. Οι, οι κανόνες του προγραμματισμού για την χωρίς ενίσχυση θα πρέπει να απλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός κανονισμού που θα εκδοθεί να γίνει πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη αυτή η διαδικασία και να επιτρέπει καλύτερη συνεργασία με τις ε, ΑΚΕ και τις ε, άκρος περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής οι, ε, τα, ΙΧΕ θα πρέπει να ε, είναι επιλέξιμες ε, για οριζοντίως για όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να απλοποιηθούν διαδικασίες που είχαμε ω τώρα. Ε, θα πρέπει να γίνουν ε, στο πρόγραμμα εργασία να συμπεριληφθούν ιδιαίτερε πρωτοβουλίε, ειδικά για τη Συχέ, γιατί ε, είναι πολύ δύσκολο στην πράξη να εκμεταλλευτούμε τι ευκαιρίε που δίδονται και θέλουμε στην πιλωτική δράση BEST ε, να συμπεριληφθεί και η βιοπικιλότητα στη ΣΥΧΕ θα πρέπει να υποστηριχθούν οι εμπορικέ στρατηγικέ των ΙΧΕ ε, θα, ε, ε, σε ό,τι αφορά τους κανόνες προέλευσης ήδη υπάρχει ένα πρωτόκολλο που δίδει προτιμησιακό καθεστώς ΙΧΕ θα τονίζουν τα συμπεράσματα αυτά τη σημασία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ε, που θα πρέπει να αναγνωριστεί ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη σημασία των υπηρεσιών αυτών για τη ΣΥΧΕ. Αυτά εισαγωγικά δίνω το λόγο στην Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ γιατί τηρήσατε το χρόνο σας, μιλώντας βέβαια με ταχύτητα φωτός. Δίνω το λόγο στον κύριο Τυρολιάν για το πρώτο πάνελ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι ο Πατρίς Τυρολιέν, ένα από τους, ένας από τους ε, τρεις εκπροσώπους της Γαλλίας που προέρχεται από τα υπερπόντια, από τις υπερπόντιες χώρες και διαμερίσματα. Από το 2009 και μετά Έχουμε και το σέμπαρτελεμί το οποίο εκπροσωπείται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ε, υπερπόντιων, ε, του σύνδεσμου υπερπόντιων χωρών και περιφερειών. Θα ήθελα να σας ε, πω ότι χαίρομαι διότι καταφέραμε να οργανώσουμε αυτή την ακρόαση και θίξαμε, μπορούμε να θίξουμε τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών και εδαφών, υπερποντίων χωρών και εδαφών. Είμαι διπλά ικανοποιημένος διότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν φύγουμε συχνά και το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζουν καλά οι ευρωβουλευτές και επίσης ε, ο χρονισμός είναι πολύ καλός διότι τώρα υπέβαλε η Κομισιόν το σχέδιό της για, που θα διέπει τις σχέσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερποντίων χωρών και εδαφών. Πιστεύω ότι θα πρέπει οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη να αποτελέσουν, να αποτελέσουν απόσπαστο μέρος της πολιτικής μας και να προβάλλουμε μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή πολιτική. Μετά από τη Συμφωνία Σύνδεσης του 2001 βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει διεθνώς τα πράγματα. Υπάρχουν νέες πολιτικές προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κλιματικές αλλαγές, περιβάλλον, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ούτω καθεξής. Και επίσης η διάρθρωση του διεθνούς εμπορίου έχει αλλάξει. Οι είχε αντιμετωπίσουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και θα πρέπει να διαθέτουν βιώσιμη οικονομία. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, διότι πρόκειται για υπερπόντιες, υπερπόντια εδάφη που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Οι είχε λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουν μία βιώσιμη οδό ανάπτυξης, αναπτύσσοντας την ανταγωνιστικότητα και μειώνοντας τον ευάλωτο χαρακτήρα των οικονομιών τους. Θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν και με τις γείτονες χώρες και ε, να βρεθούν στο παγκόσμιο προσκήνιο. Θα πρέπει να ορίσουμε μια σωστή πλαισίωση ανάπτυξης των είχε. Βλέπουμε ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η είχε προωθούν μια νέα βάση συνεργασίας η οποία προσαρμόζεται καλύτερα στα διεθνή πλαίσια, δηλαδή μείωση της φτώχειας, καλύτερη εταιρική σχέση, ενισχυμένη οικονομική εταιρική σχέση για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, ε, προστασία του περιβάλλοντος, αξιολόγηση της βιοποικιλότητας και ανάπτυξη του εμπορίου και του τουρισμού. Αυτοί είναι οι πυλώνες τους οποίους βασιζόμαστε για να φτάσουμε σε μια σωστή εταιρική σχέση. Σε σχέση με την αξιοποίηση της βιοπικιλότητας που διέπει της είχε, έχουμε τα νέα προγράμματα ε, live και προβλέπονται νέα σχέδια και προγράμματα η Επιτροπή δεν επιτρέπει στα, στις ΙΧΕ να προβάλλουν σχέδια και προγράμματα τα οποία να κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από, τα, από τις υπερπόντιες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Γενική Διεύθυνση του Περιβάλλοντος όμως να τηρήσει στο ακέραιο της υποχρεώσης της. Ξέρουμε ότι οι εμπορικές σχέσεις είναι πρωταρχικής ε, σημασίας για να μπορεί κανείς να είναι αυτόνομος στο εμπορικό προσκήνιο. Γι' αυτό και η πρόταση σύνδεσης ενέχει ορισμένες αντιφάσεις. Υπάρχουν νέες διαδικασίες πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις των ΙΧΕ που θέλουν να εξάγουν προς τις ευρωπαϊκές χώρες και αυτές οι νέες ε, διατάξεις δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί στην ελεύθερη αγορά. Χρειάζεται ένα σημαντικός χρόνος προσαρμογής για τις είχε, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Τέλος, η Επιτροπή δεν εξετάζει επαρκώς τους κανόνες προέλευσης και οι επιχειρήσεις των ΙΧΕ δεν έχουν ε, επαρκή πρόσβαση. Αυτό αφορά τον Μαυρίκιο και τις Σεϊχέλες ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ. Δυστυχώς ε, δεν υπάρχει ε, πλήρης διαφάνεια μέσα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας σύνδεσης με τις ΙΧΕ. αφήσω, θα δώσω το λόγο στους παρεμβαίνοντας του πρώτου πάνελ για να μας παρουσιάσουν τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας στα υπερπόντια εδάφη και χώρες για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε την αυτόχθονη ανάπτυξη. Δεν ξέρω ποιος θα λάβει το λόγο πρώτος. Oui, oui, à Monsieur Gaston et... Euh, Ο κύριος Γκαστόν, οι κύριοι Γκαστόν και Βάλ έχουν το λόγο. Μπορώ να μείνω εδώ για να, έχω, να κάνω την παρουσίασή μου, όπως επιθυμείτε. Θα ακούσετε τον κύριο Γκαστόν, Ολιβιέ Γκαστόν, που αντιπροσωπεύει ε, την Σέμπιαρ ε, και Μικλόν στο Παρίσι είναι αντιπρόεδρος της ε, Ένωσης ε, ΙΧΕ. Donc, monsieur, monsieur Gaston, d'abord, Ευχαριστώ κύριε Τυρολιά, κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Ολιβιά Γκαστό. Προσθέτω, όπως είπε και η Κλώη Κλαβινιάκ, ότι η Πιέρ και Μικλόν θα αναλάβει την Προεδρία της Ένωσης ΥΧΕ από την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι λοιπόν πολιτικός συνομιλητής την επόμενη χρονιά μαζί με και δίπλα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ε, Ένωσης ΥΧΕ της Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε τους ε, τρεις συνδιοργανωτές, ευρωβουλευτές. Ε, το αντικείμενο για το οποίο θα μιλήσω είναι οι ανταγωνιστικές είχε για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Πράγματι, η ανταγωνιστικότητα είναι ένας από τους στόχους της ε, απόφασης ε, σύνδεσης. Η παρέμβαση μου θα έχει τρία τμήματα. Πρώτον, θα μιλήσω για το περιβάλλον ε, και για τα του, για τα πλεονεκτήματα των ΙΧΕ. Δεύτερον, πώς μπορούν οι ΙΧΕ να γίνουν ανταγωνιστικές στο πλαίσιο ε, της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Και τρίτον, τι μπορεί να γίνει σήμερα με την αναθεώρηση της απόφασης σύνδεσης. Λοιπόν, νομίζω ότι η προηγούμενη ομιλητές ε, έθεσαν τη βάση, ε, το, το, μας εξέθεσαν το περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι χέ, πληθυσμός, έκταση κλπ. Εγώ θα ε, σταθώ πιο πολύ στα πλεονεκτήματά τους που βοηθάνε τις ΧΕ να είναι πιο ανταγωνιστικές αλλά είναι πλεονεκτήματα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναπτυξιακή της πολιτική. Πρώτο πλεονέκτημα η βιοπικιλότητα. Δεν θα επιμείνω πολύ, διότι ε, σε λίγο θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτήν. Είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τη ΣΥΧΕ. Περίπου το 90% της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας εκτιμάται ότι βρίσκεται σε υπερπόντια, ε, υπερπόντιες περιοχές, κυρίως χώρες και εδάφη. Δεύτερον, φυσικός πλούτος που πολύ συχνά βρίσκεται στο κέντρο των ιστορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη ΣΥΧΕ. Αποτελεί επίσης και αντικείμενο της Συμφωνίας Αλληλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Γρυλανδίας. Βλέπετε τι τύπους ε, συνεργασίας, ε, ποιοι τύποι συνεργασίας είναι κοινού συμφέροντος. Η Νέα Καλλιδονία, για παράδειγμα, ε, είναι πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους. Ε, μετά, οικονομικές, ζώνε ε, οικονομικές ζώνες αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Την Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία ε, έχουν το περισσότερο από 85% των ζωνών αυτών υπερπόντια. Η Γαλλία, για την ακρίβεια, ε, έχει μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες την ε, δεύτερη σε μέγεθος ε, νησιωτική οικονομική ζώνη στον κόσμο. Αυτό συνδέεται βέβαια και με τους φυσικούς πόρους αλλά και με τον τουρισμό ο οποίος επίσης είναι πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας ε, στη ΣΥΧΕ. Υπάρχουν δύο μοντέλα ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στη ΣΥΧΕ. Πρώτον, που βασίζεται, ένα μοντέλο που βασίζεται στο φυσικό πλούτο και το δεύτερο μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται πιο πολύ σε, επιχειρήσεις προς τις, ε, ε, σε υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και τουρισμό πολυτελείας. Αυτό είναι το μοντέλο πιο πολύ δουλεύει αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι αυτού, αυτού του είδους τα μοντέλα είναι δύσκολο να αντιγραφούν σε άλλες περιοχές ε, και αυτό ισχύει και για τους φυσικούς πόρους ε, και για το δεύτερο μοντέλο και ιδιαίτερα για τους φυσικούς πόρους υπάρχει ένα, φυσικούς πόρους είναι, υπάρχει ένα θέμα βιωσιμότητας γιατί βέβαια φυσικοί πόροι εξαντλούνται κάποια στιγμή θα πρέπει σε συνάρτηση με το περιβάλλον τους ε, η, η, η, κάθε ηχέ να βρει το δικό της μοντέλο για παράδειγμα, ε, να λαμβάνοντα υπόψη την πράσινη ανάπτυξη με διάφορα project όπως ε, στην Αρούμπα που έχει ένα πολύ φιλόδοξο ενεργειακό πρόγραμμα, ε, στις Μαλβίνες που έχουν ένα πολύ προχωρημένο σύστημα διαχείριση των ελευτικών της πόρων ή σε οποιαδήποτε άλλη είχε που θέλει να εφαρμόσει την πράσινη ανάπτυξη με άλλα project. Πώ η ανταγωνιστικότητα θα μπει στην υπηρεσία της βιώσιμη ανάπτυξη, Σε αυτή τη διαφάνεια ε, βλέπουμε το πώ συνδέονται οι τρει ε, ε, στόχοι του σχεδίου απόφαση σύνδεση, του οποίου υπενθύμισε ο κ. Τυρολία αυξημένη ανταγωνιστικότητα πάνω αριστερά, μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογή, πάνω δεξιά και μεγαλύτερη συνεργασία και περιφερειακή ολοκλήρωση κάτω. Δεν θα μιλήσω με λεπτομέρειε για αυτά, αλλά είναι σαφές ότι η ανταγωνιστικότητα υποστηρίζει τους δύο άλλου στόχου. Γιατί η αυξημένη ανταγωνιστικότητα καθιστά τις περιοχές αυτές ε, πιο ανθεκτικές σε οποιαδήποτε, ε, οποιαδήποτε κρίση και σοκ, ε, οικονομικό, περιβαλλοντικό κλπ. Και ταυτόχρονα επιτρέπει την μεγαλύτερη ολοκλήρωση περιφερειακή και τοπική. Βέβαια ισχύει και το αντίστροφο, η μεγαλύτερη ολοκλήρωση αυξάνει την ανταγωνιστικότητα. Μετά, ας δούμε πώς μπορούμε να συμφιλειώσουμε την ε, πολιτική ανταγωνιστικότητα με την βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει ένα ε, αναπτυξιακό εργαλείο πολύ χρήσιμο, ε, το οποίο άρχισε να χρησιμοποιείται από την πρώτη διάσκεψη του Ρίο πριν από 20 χρόνια είναι η Ατζέντα 21. Ατζέντα σημαίνει τι πρέπει να γίνει. Ε, είναι ένα πρόγραμμα δράσης δηλαδή που θα επιτρέψει να ασκηθεί μια κρατική πολιτική υπέρ τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε διάφορα επίπεδα. Το 90% τη Ατζέντα 21 αυτή τη στιγμή ε, εφαρμόζεται στην Ευρώπη με ελάχιστε εμπειρίες σε ΙΧΕ. Ε, ποια είναι τα διδάγματα από την Ατζέντα 21, οι στόχοι τη ε, για την ακρίβεια, η, πρώτον η συμμετοχή, η συμμετοχή όλων των οικονομικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών φορέων κλπ. που θα επιτρέψει όχι μόνο να ληφθούν υπόψη οι εμπειρίες τους, αλλά και να γίνουν ε, πομπή της περιφερειακής πολιτικής. Ε, δεύτερον, ε, αντί να έχουμε τομεακές πολιτικές περιβάλλοντος ή ανταγωνιστικότητας, η Ατζέντα 21 θα επιτρέψει, επιτρέπει τη σύνδεση αυτών. Επίσης δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση. Γιατί η αξιολόγηση θα επιτρέψει η βοήθεια να γίνει πιο αποτελεσματική και να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα με τέτοια ποσά. Ε, η Ατζέντα 21 στις ΙΧΕ ε, εντοπίζεται πιο πολύ στην Γουαδελούπη ε, και αλλού σε άκρος περιφερειακές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή στην Κουάουα επίσης όπου έχουμε ένα πρώτο πείραμα και κάποια άλλα τα οποία θα ξεκινήσουν Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε λοιπόν τη σημασία αυτού του εργαλείου στις ΙΧΕ. Ποιοι είναι οι παράγοντες ανταγωνιστικότητας που θα επιτρέψουν στις ΙΧΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ε ενισχύσουν την ανάπτυξη των ΙΧΕ. Ε, καταρχήν, τοπικοί παράγοντες, φυσικός ε, πλούτος, ε, περιφερειακή ολοκλήρωση, προσβασιμότητα. Προσβασιμότητα σημαίνει επενδύσεις στις υποδομές που θα συνδέσουν τη συχεία με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, το επιχειρηματικό περιβάλλον, ο χρόνος για παράδειγμα δημιουργίας μιας επιχείρησης περνάει από μία μέρα σε ορισμένες είχε σε έξι μήνες σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής στις είχε το διάστημα αυτό είναι από μερικέ μέρε μέχρι μερικέ εβδομάδε, αυτό είναι ο μέσο όρο. Ε, Επίση είναι πολύ σημαντική τεχνολογία, ε, ανθρώπινο, το ανθρώπινο δυναμικό και η επιστημονική προσέγγιση. Βλέπουμε ότι η στρατηγική των πόλων ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσει είναι μια στρατηγική πετυχημένη. Είναι μια αναπτυξιακή στρατηγική που υποστηρίζεται όλο και περισσότερο στη ΣΥΧΕ. Επίσης υπάρχουν και διεθνεί παράγοντες. Έχουμε μιλήσει για την εμπορική πτυχή της Συμφωνίας Σύνδεσης με τη ΣΥΧΕ. Η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι πολύ σημαντική και σε ό,τι αφορά την ε, τους κανόνες προέλευσης όσο και την προτιμησιακή πρόσβαση. Μπορείτε να διαβάσετε την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Εμπορίου που ακριβώς σχολιάζει αυτούς τους παράγοντες ε, που είναι πολύ σημαντικοί στις εμπορικές σχέσεις, ε, συμφωνίες. Συγγνώμη. Τι μπορεί να γίνει τι μπορεί να γίνει σήμερα στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης. Ας δούμε τι έγινε στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης. Είχε Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ε, είπε η ΚΛΟΕ, έχει προσθέσει ε, πραγματική αξία στη σχέση, έχει προσθέμενη αξία αυτή η σύνδεση, αυτή η σχέση. Έχουμε τους ε, την ενίσχυση η οποία επιτρέπει στη ΙΧΕ να ε, ενισχύσουν την παγκληματική κατάρτιση, την εκπαίδευση, της ε, υποδομές. Αυτό σε τοπικό επίπεδο. Μετά σε περιφερειακό επίπεδο η ενισχύση και η σχέση αυτή επέτρεψε την εκπόνηση στρατηγικών καινοτομία ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπω για παράδειγμα στην Καραϊβική. ή ε, έχει δοθεί χωρί δασμού πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά από πλευρά των ΙΧΕ και οι κανόνες ε, ε, προέλευσης επίσης βοηθούν πάρα πολύ τι ΙΧΕ δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Τώρα, τι, μπορεί να γίνει παραπάνω μπορεί να γίνει με το σχέδιο αποφάσης για ε, σύνδεση το οποίο συζητούμε. Καταρχήν, η διατήρηση της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την προηγούμενη απόφαση, η ενίσχυση που δόθηκε προς τη Συχία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 1,7% του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Θα πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη και τα, τα συμφέροντα των ΙΧΕ όταν υπογράφονται εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Όταν συνάπτονται συμφωνίες όπως για παράδειγμα με τις χώρες ΑΚΕ ε, ή με τον Καναδά, οι ΙΧΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη γιατί αυτές οι χώρες, Καναδάς για παράδειγμα, χώρες ΑΚΕ, είναι γειτονικές των ΙΧΕ η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου με τρίτες χώρες επηρεάζει την οικονομία, τις οικονομίες των ΙΧΕ, γιατί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επαφής με αυτές τις χώρες με τις οποίες συνάπτονται συμφωνίες απελευθέρωση του εμπορίου. Επίσης, ό,τι αφορά τους κανόνες προέλευσης, ε, μιλήσαμε ε, για το ε, πιο προνομίουχο καθεστώς, Το καταλαβαίνουμε πολύ στον τομέα των υπηρεσιών, όμως στον τομέα των αγαθών οι κανόνες προέλευσης μερικές φορές είναι πιο προτιμησιακοί, πιο ευνοϊκοί μάλλον να το πω έτσι, για ορισμένες χώρες και δεν χορηγείται το καθεστώς του ε, πιο ε, ευνοούμενου ε, κράτους της ΙΧΕ. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία της ε, ανταγωνιστικότητας ε, που είναι, οικονομικός, ε, που είναι πολύ σημαντικός παράγων για την οικονομία. Τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε από το σχέδιο απόφασης ε, θέλουμε ε, να ε, ενταχθούν περισσότερο οι, ΙΧΕ ΧΕ στις διαπραγματεύσεις με συμφωνιών για με τρίτες χώρες, να διευρυνθεί ο χαρακτήρας του πιο ευνοούμενου κράτους που χορηγείται στις ΙΧΕ και επίσης ορισμένοι οικονομικοί τομείς να ενταχθούν στο στο συνολικό κεφάλαιο της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έτσι ώστε να, γίνει, να μπορεί να ε, γίνει συνεργασία και σε αυτούς τους τομείς. Ε, η, ΧΕ, η σχέση με τις ΙΧΕ πραγματικά θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνδυασμό της ανταγωνιστικότητας με την βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος... Μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής δυστυχώς. Ο κύριος Τυρολιέν χωρίς μικρόφωνο, επόμενος ομιλητής, θα πάρει το λόγο. Euh, euh, Καλημέρα σας. Θα κάνω την παρουσίασή μου στα αγγλικά. Θα πρέπει να σας ε, δώσω εξηγήσεις για ένα τεχνικό, τεχνικής υφής ε, ζήτημα σε μια άλλη γλώσσα από αυτή που ακούστηκε μέχρι τώρα. Η παρουσίασή μου έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα, με την βιώσιμη ανάπτυξη και με την ανθεκτικότητα αυτών των υπερποντιών χωρών και, με, και τι μπορεί να συνεισφέρει αυτή η απόφαση σύνδεσης στον τομέα του εμπορίου. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, στα επόμενα δέκα λεπτά θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το νεότερο σκεπτικό της ε, Κομισιόν για το πώς το εμπόριο μπορεί να συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα, την βιώσιμη ανάπτυξη και την αντακτικότητα. Θα το βρείτε στην πρόταση του Ιουλίου, αλλά σήμερα αυτά που θεωρούμε εμείς τις τρεις μεγάλες ε, κοινοτομίες ε, στον τομέα της συνεργασίας θα τις παρουσιάσω ενώπιον σας. Καταρχάς, ενισχυμένες ε, συνθήκες για εξαγωγές στις, ε, στα υπερπόντια εδάφη, έπειτα βελτιωμένη πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες των ΙΧΕ και τρίτον καλύτερο, καλύτερη εστίαση στα ζητήματα εμπορίου και συνεργασίας. Ονομάζομαι Ρέμ Κοβάλ, είμαι αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ασχολούμαστε με τις συμφωνίες ε, εμπορικής συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ, αλλά και επίσης με την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς τις χώρες ΙΧΕ. Δεν είμαι και εμπειρογνώμονα για τα πάντα που έχουν σχέση με τις υπερπόντιες χώρες, διότι θα χρειαστεί μια ολόκληρη ζωή για να τα μάθει κανείς όλα. Δεν θα σας μιλήσω προς το παρόν για τις προπαρασκευαστικές εργασίες, διότι τα έγγραφα είναι δημόσια και μπορείτε όλοι να τα διαβάσετε αν επιθυμείτε. Θα προχωρήσω άμεσα στις τρεις αυτές καινοτομίες που ανέφερα όσον αφορά τα εμπορεύσιμα αγαθά. Δεν ήταν εύκολη η καινοτομία. Και γιατί? Διότι η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει το, καθεστώς, το εμπορικό καθεστώς και οι υπερπόντιες χώρες λαμβάνουν αφορολόγητα, αφορολόγητη πρόσβαση και χωρίς ποσοστώσεις. Και πώς μπορεί όμως αυτό να βελτιωθεί. Ε, εμείς θεωρήσαμε αναγκαίο ε, δεδομένου ότι η απόφαση, η σχετική απόφαση είναι πάνω από 10 ετών. Με λίγα λόγια προτείναμε τρία διαφορετικά πράγματα. Καταρχάς, να εξυγχρονίσουμε και να βελτιώσουμε τους κανόνες που καθορίζουν πώς μπορούν να, να επωφεληθούν οι υπερπόντιες χώρες από την πρόσβαση αυτή. Έπειτα, να καθορίσουμε συγκεκριμένους κανόνες που θα διευκολύνουν την ομαλότερη πρόσβαση τις ε, περιπτώσεις επίσης όπου θα χρειαστεί να αρνηθεί η πρόσβαση και τρίτον να ζητήσουμε από τις υπερπόντιες χώρες να μην κάνουν διακρίσεις εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα ε, και προς αναδυόμενες οικονομίες όπως την Ινδία ή την Κίνα. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ίσως ακούσατε ήδη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει αυτούς τους ε, κανόνες. Μέσα στα 10 χρόνια που ισχύουν αυτοί οι κανόνες έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Υπάρχει το σύστημα GSP, στο οποίο θα βρείτε τους πιο σύγχρονους κανόνες. Και αυτοί αποτέλεσαν την βάση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κανόνες πρέπει να απλοποιηθούν, να γίνουν πιο χαλαροί, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ε, αλλιευτικά προϊόντα και το παράδειγμα που θα σας δώσω είναι ο κανόνας που καθορίζει τον προσδιορισμό της εθνικότητας ενός αλλιευτικού σκάφου και τις προδιαγραφές εθνικότητας για το πλήρωμα του πλοίου αυτού. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να απαλληφούν αυτές οι προδιαγραφές έτσι ώστε τα αλλιευτικά προϊόντα να λάβουν ε, χώρα προέλευσης ε, υπερποντίων εδαφών. Επίσης, πιστοποίηση προέλευσης από καταγεγραμμένους εξαγωγείς. Στην περίπτωση αυτή, οι ίδιοι εξαγωγείς θα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν την προέλευση των προϊόντων τους. Αυτό απαιτεί μία μεταβατική περίοδο όπως είπε και ο κύριος Τιγαουλιά, θα αρχίσει το 2017. Στόχος όμως είναι να απλοποιηθούν οι εξαγωγές. Θα παραμείνω σε αυτόν τον τεχνικό τομέα, διότι προτείνουμε και βελτιώσεις στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, στο GSP. Θα αναφέρω τρεις από αυτούς. Καταρχάς, την απλοποίηση, την περαιτέρω απλοποίηση της πιστοποίηση προέλευση, το οποίο θα υποφελήσει τις ε, μικρές, πολύ μικρές περιφέρειες, έπειτα να επικαιροποιηθούν να επικαιροποιηθεί η δυνατότητα ε, παρέκκλησης το σύστημα αυτό, το χρονικό περιθώριο των 5 ετών, έτσι ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις ανάλογα με την περίπτωση. Τέλος, η προέλευση. που θα διευκολύνει την συμμόρφωση με τους κανόνες την χώρα προέλευσης. Επίσης, περιορίζει τις ε, δεν θα περιορίζει τις ε, δυνατότητες πρόσβασης της χώρας ΑΚΕ και, τις, ε, και τα περπόντια εδάφη. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε τον κανονισμό αυτό πέρα από τις υπερπόντιες χώρες σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν ολοκληρώσει είτε συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας είτε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε που λαμβάνουν ένα ειδικό προτιμησιακό καθεστώς και αυτό θα διευρύνει την ομάδα αυτή των χωρών. Φυσικά πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις έτσι ώστε να, οι χώρες αυτές να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους αυτό το ειδικό καθεστώς. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δείτε ότι παρέχει πολλές ευέλικτες δυνατότητες. Αυτά εν ολίγης για τους κανόνες προέλευσης. Στη, στη δεύτερη και την τρίτη καινοτομία θα είμαι λίγο πιο σύντομο. Πρώτον για τις υπηρεσίες, εμπορικές υπηρεσίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίε είναι πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο των οικονομιών των χωρών αυτών. Είναι η ραχοκοκαλιά τη σύγχρονη οικονομία, η ραχοκοκαλιά των ανταγωνιστικών ε, εξαγωγών. Η παρούσα απόφαση πάλι χρονολογείται πάνω από 10 έτη. Υπάγεται στον, στον ΠΟΕ και αυτό σημαίνει ότι τα υπερπόντια εδάφη ε, αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΠΟΕ. Και από τότε που δημιουργήθηκε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένε Πολιτείε μέσω διμερών συμφωνιών άρχισαν να προσφέρουν καλύτερους εμπορικούς όρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι τα υπερπόντια εδάφη πρέπει να απολαμβάνουν πολύ καλύτερης μεταχείρισης ε, κατά από αυτή την απόφαση και κάτι άλλο που εντοπίσαμε είναι η διάταξη του, της πιο αγαπημένης χώρας, όπως λέγεται, η χώρα δηλαδή που αυτόματα θα λάβει την καλύτερη μεταχείριση ή που έλαβε στο παρελθόν ή που θα λάβει στο μέλλον. Και το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη δυνατή μεταχείριση για αυτές τις ευνοούμενες χώρες που είπε και ο κύριος Σαραμαντής οι δεσμεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υπηρεσίε αυτές θα είναι πολύ πιο φιλελεύθερες από ό,τι τώρα και θα συνεισφέρουν στην δημιουργία νέων συμφωνιών ακόμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχω να σας πω σήμερα. Τρίτη καινοτομία τον τομέα της ε, συνεργασίας και των εμπορικών ζητημάτων. Καμία εμπορική συναλλαγή δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την συνεργασία και χωρίς ε, προδιαγραφές που ευνοούν και διευκολύνουν αυτήν την συνεργασία στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Η τωρινή απόφαση περιλαμβάνει ε, διάφορες προδιαγραφές, υγειονομικές προδιαγραφές από αυτές μέχρι ανταγωνιστική πολιτική. Θα βρείτε και εδώ τι λεπτομέρειε στην πρόταση τη Κομισιόν. Και τι κάνει η Κομισιόν με αυτή την πρόταση, τρία πράγματα. Επικαιροποιεί τι τις ε, ισχύουσε διατάξει έτσι ώστε να ενδυναμώσει τι δυνατότητε των υπερπόντιων χωρών και να συνεισφέρει σε ένα καλύτερο επιχειρηματικό κλίμα, όπω ήδη αναφέρθηκε από τον κύριο Γκαστό είναι τα κύρια συστατικά στοιχεία της καλής οικονομίας ή βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα και προδιαγραφές σχετικές με την φορολόγηση, έτσι ώστε να προωθηθεί η χρηστή διακυβέρνηση στις περιοχές κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπερπόντιες ε, χώρες και εδάφη. Αυτά για, τα, για τη συνεργασία μας στα εμπορικά ζητήματα. Εμείς προτείνουμε έναν διάλογο για συνεργασία και να δώσουμε, να εστιάσουμε στην, ε, να εστιάσουμε καλύτερα στην οικονομική συνεργασία από ό,τι στο παρελθόν. Τελειώνω με ένα σύντομο συμπέρασμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε τρία κύρια εμπορικά στοιχεία για να προωθήσει τους τρεις αυτούς στόχους Οι κανόνες προέλευσης στα εμπορικά αγαθά, οι ευνοούμενες χώρες στις εμπορικές συναλλαγές και στις επενδύσεις και ο καλύτερος διάλογος για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ τους παρεμβαίνοντες. Λέει ο κύριος Τυρολιά. Προβέλεπετε λοιπόν ανταλλαγή απόψεων. Βλέπω όμως ότι δεν είναι και τόσο αθρώα η προσέλευση. Δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Δεν ξέρω τι διάσταση θα έχει. Τι διαστάση θα έχει θα ήθελε να λάβει κάποιο το λόγο για να υποβάλει ερωτήσεις προς το πάνελ. Η κυρία Θεοχάρους. Κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις θα ήθελα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να απαντήσει. Βεβαίως σας συγχαίρω για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και ακούσαμε πολλά στοιχεία που λίγος πολύ απασχολούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα απομακρυσμένα νησιωτικά κράτη και το κεντρικό πυρήνα και τις ε, ε, υπερπόντιες χώρες. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που μια περιοχή θελήσει να πάρει την αποκλειστική οικονομική της ζώνη και να φύγει, να αυτονομηθεί, να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Ποια θα είναι η σύνδεση τη από εκεί και πέρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο καθεστώς έχουν οι πολίτες της χώρας αυτής, οι οποίοι τώρα είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Και απ' την άλλη, αν μια περιοχή θελήσει να αποκτήσει αυτό το καθεστώς, γιατί στην άμεση γυτνίαση υπάρχουν και άλλα ανάλογα περιστατικά. Ξέρω την, την περίπτωση της στην Καραϊβική. Τι θα συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Τέλος ήθελα να ρωτήσω ποιες περιοχές έχει το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι υπερπόντια εδάφη με αυτό το καθεστώς. Για παράδειγμα, ε, συγχωρέστε μου την άγνοια, αλλά το Γιβραλτάρ τι καθεστώς έχει. Οι στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο τι καθεστώς έχουν. Τα Φόκλαντς, ε, το, η Σεντελίνα. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να έχω μια πληροφόρηση, γιατί τις προάλλες άκουσα και τον συνάδελφό μας, τον κύριο Γκάραχμ, να λέει ότι εκλέγεται από τους κατοίκου του Γιβραλτάρ. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κάποιες ε, συγχύσει. Και γιατί δεν έχουμε ούτε ένα ευρωβουλευτή από την Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, να ακούσουμε και εκείνον την άποψη. Ευχαριστώ. E, e, za i za informacje, które Σας ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Πράγματι, το πρόβλημα, το θέμα αυτό μας απασχολεί διότι και η Επιτροπή Ανάπτυξης θα υποβάλει μια εκθέση επί του θέματος. Γι' αυτό αυτή η ακρόαση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, θεωρώ. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση σε σχέση με την συνεργασία των τεσσάρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με τις υπερπόντιες χώρες. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται, τι έγινε μάλλον με τη συνεδρίαση των ε, ΑΚΕ στη Δανία. Είδαμε ότι υπάρχει και θέμα ε, ε ανεξάρτητας ανεξαρτησίας, με συγχωρείτε, στο μέτρο της ενέργειας. Δηλαδή, ορισμένες χώρες θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν στον τομέα της ενέργειας. Είναι θέμα επικαιρότητα και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτές οι εμπειρίες θα πρέπει κάτι να μας διδάξουν, διότι η Δανία είναι προτεργάτη ε, στον τομέα της ενέργειας και στις ανανεώσιμες. Ο κύριος Παλαζή, ένα ερώτημα τεχνικής υφής που έχει σχέση με το εμπόριο. Μιλήσαμε για τη βιοπικιλότητα που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των είχε και μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με το εμπόριο και επειδή μιλάμε για είδη τα οποία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα, θα πρέπει να δούμε πώς ε, γίνονται έλεγχοι στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, διότι υπάρχουν ε, ήδη ενισαγωγοί που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα. Θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι όπως στην Αυστραλία και στη Ισλανδία, διότι εκεί υπάρχει μεγάλος έλεγχος. Στην Ταϊτή υπάρχει ένα είδος που λέγεται μικόνια, και το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί και να εξαχθεί προς τα έξω. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενεχόμενο στόχος και οι νίκητες και τα διάφορα φυτά όταν εισαχθούν σε μια χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξαλειφθούν. Θα ήθελα λοιπόν η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να λάβει υπόψη αυτή τη διάσταση γιατί και οι είχε θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτές τις εισαγωγές ε, οι οποίες μετά δεν μπορούν να αφορούν ήδη που δεν μπορούν να εξαλειφθούν. σε σχέση με το ερώτημα που θίξατε, που έθιξε η κυρία Θεοχάρους, τι θα γίνει με την ενδεχόμενη ανεξαρτησία ορισμένων χωρών, εγώ μπορώ να απαντήσω μόνο για τις είχε που σχετίζονται με τη Γαλλία. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω μόνο για την περίπτωση της Γαλλίας. Το άρθρο 73 ή 74 του συντάγματος επιτρέπει σε ορισμένα συμπλέγματα να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους, αν το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει και για τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα. Υπάρχει η δυνατότητα να περάσει κανείς από υπερπόντιο διάρισμα, διαμέρισμα να περάσει από αυτό το καθεστώς στην ανεξάρτητη χώρα. Το, ο Άγιος Βαρθολομέος, το Σεν έχει ε, αλλάξει καθεστώς και θεωρείται τώρα είχε. Θα μπορούσε να ισχύσει και η αντίστροφη πορεία, δηλαδή στο Σεν Πιέρε Μικλόν, για παράδειγμα, το 2014 θα γίνει μία υπερ-απομακρυσμένη περιφέρεια. Ο, η, η νήσι Μικλών ήταν πετεών, δηλαδή είχε μέχρι τούδε. Και στη συνέχεια μπορούν ε, να αλλάξουν καθεστώς και να θεωρηθούν υπερπόντια διαμερίσματα. Μετά μπορούν να ξαναλλάξουν καθεστώς αν το επιθυμούν. Όλα εξαρτώνται από την διάθεση αυτών των κρατών και από το Σύνταγμά μας. Αυτά τα υπερπόντια εδάφη μπορούν να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους. Εάν το ε, επιθυμούν εγώ, προέρχομαι από τη Γουαδελούπη, η οποία κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ανεξάρτητη χώρα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και το προβλέπει και το Γαλλικό Σύνταγμα. Δηλαδή, μία πλέον απομακρυσμένη περιφέρειά μας μπορεί να κηρύξει την ανεξαρτησία του. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά προβλέπεται από το Γαλλικό Σύνταγμα. Το ίδιο ισχύει και για ένα υπερπόντιο διαμέρισμα το οποίο μπορεί να κηρύξει την ανεξαρτησία του. Δεν ξέρω τι ισχύει στις άλλες χώρες οι διαμερίσματα και τι ορίζουν τα άλλα τρία κράτη εάν ε, διαβλέπετε, αν προβλέπετε αυτή η δυνατότητα, για τις άλλες χώρες δεν μπορώ να ε, αποφανθώ. Αλλά στην περίπτωση της Γαλλίας προβλέπετε αυτή η δυνατότητα από το Σύνταγμά μας. Αν μου επιτρέπετε να δώσω κι εγώ κάποια πιο συγκεκριμένα ε, πρόσθετα στοιχεία, το πέμπτο τμήμα της πρότασης της Κομισιόν προβλέπει την περίπτωση το Συμβούλιο να αποφασίσει προσαρμογή της ε, απόφασης σύνδεσης όταν ε, στις εξής περιπτώσεις. Πρώτον, ένα, μία είχε γίνεται ανεξάρτητη, ανεξάρτητο κράτο. και εγκαταλείπει την Ένωση. Το, η απόφαση του Συμβουλίου του 2001 αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε τέτοιου είδου περίπτωση. Ε, δεν εφαρμόζεται για τις Βερμούδες επειδή ε, το επέλεξαν. Όμως η οι Βερμούδες ε, είναι στον κατάλογο ηχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η απόφαση σύνδεση του 2001 δεν εφαρμόζεται στις Βερμούδες. επόμενη περίπτωση όταν μια ηχεία γίνεται άκρος περιφερειακή περιοχή ή το αντίστροφο. Σε, μία από αυτές, σε οποιαδήποτε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί το Συμβούλιο να αποφασίσει την προσαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Σε ό,τι αφορά την λίστα των ηχέ, το παράρτημα 2 της Συνθήκης απαριθμεί όλες αυτές τις ηχέ σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν 12 ε, ε, είχε το Γιβλαρτάρ δεν και, και οι βάσεις στην Κύπρο δεν συμπεριλαμβάνονται όμως υπάρχουν ηχές στην Καραϊβική την, η Αγκουίλα, οι Βερμούδες ε, η νησί Κάιμαν Μονσεράτ Τέρξεν Κέικος Βέβαια, η νήσι Φόκλαντ, η Αγία Ελένη και στον Ανταρκτικό έχουμε την, ε, Βρετανικές, ε, ε, τη Βρετανική, Βρετανικές Στην, όμως το παράδειγμα 2 της συνθήκης απαριθμεί πραγματικά εξαντλητικά όλες τις ηχέ. Με απόφαση του Συμβουλίου τροποποιήθηκε για να προσθεθεί ο Άγιος Βαρθολομαίος από 1η Ιανουαρίου 2012, απόφαση του, Συμβουλίου που, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που οδήγησε το, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ε, τροποποιήσει την απόφαση του 2001 έτσι ώστε να ε, λάβει υπόψη της, ε, την συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αλλαγή της συνθήκης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους δύο επόμενους ε, ομιλητές, ε, το κύριο, τους κυρίους Ιβριάν και Παλαζή. Σας παρακαλώ να έρθετε εδώ για το δεύτερο τμήμα της ακρόασης αυτής. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Ζακί Μπριγιάν. Ο κύριος Ζακί Μπριγιάν μας επισκέφτηκε κατά το φόρουμ των είχε στο παρελθόν. Είναι ένας νέος υπουργός, ο οποίος άρχισε τη σταδιοδρομία του στην Μπόρα Μπόρα, ήταν διευθυντής σχολείου και συνεργάζεται μακρόν μαζί μας ασχολείται με τις πυρηνικές δοκιμές στον Ειρηνικό και εκείνος ε, ήταν ο πρωτοστάτης αντιμετώπισης των πυρηνικών ε, δοκιμών στην Πολυνησία και είναι Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας ε, και Ορυχείων. και ίσως γνωρίζετε ότι ασχολείται και με πολιτισμικά ζητήματα. Εγώ τον γνωρίζω και υπ' αυτή του την ιδιότητα. Θα μας μιλήσει για την αηφόρο ανάπτυξη. Θα μας μιλήσει για την ε, πράσινη ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι είχε υπόκεινται σε κλιματικές αλλαγές και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια στρατηγική θα εκπονήσουν τα υπερπόντια εδάφη για να επιβιώσουν. Αυτό το ερώτημα είχα θέσει στον κύριο Μπρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναθέσει θέση μελέτες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικές καταστροφές, κλιματικές αλλαγές, απειλές για τη βιοποικιλότητα, παράνομη αλληλεία, απόβλητα. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ζακή Μπρία, ε, θεωρείται ως Υπουργός Περιβάλλοντος ότι αυτές οι προτεραιότητες επαρκούν. Στις δικές μας χώρες Οκενίας και του Ειρηνικού ε, λέμε Γιωράν. Ζητώ συγγνώμη από τους μεταφραστές, είναι λίγο δύσκολη η λέξη αυτή να μεταφραστεί. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, συνδιοργανωτές γιατί μας δίνουν ένα βήμα να εκφράσουμε τη σκέψη μας. Πράγματι, στην εισαγωγική σας παρουσίαση θα ήθελα... Α, να πω ότι με συνοδεύει ο Λιβέ Σαμπιόν που είναι διευθυντής του πολιτικού γραφείου. Ε, κλείνει παρένθεση. Υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό που είναι το πολιτιστικό για τον Ειρηνικό ωκεανό. Ε, και γιατί ε, η ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πολιτιστικό στοιχείο. Αυτό δεν το λέω για να προσθέσω λίγο folklore στη συζήτηση. Ούτε επειδή είναι της μόδας ε, να διεκδικεί ο καθένας την πολιτιστική του ταυτότητα ή την διαχείριση των πόρων του. Θα σας δείξω μια, θα σας δώσω μια εξήγηση μέσω της ε, δικής μας κουλτούρας και της γλώσσας μας. Δυστυχώς μιλάει χωρίς μικρόφωνο τώρα. Αυτό το τραγούδι είναι χαρακτηριστικό όταν οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας ε, έφευγαν για τη θάλασσα να πάνε να ψαρέψουν. Ε, και ευχαριστούσαν τον ε, καιρό ε, τον ουρανό ε, για τον καλό καιρό που θα τους έδινε. Είναι κάτι πολύ παλιό. Σήμερα εξακολουθούμε να μιλάμε για συμβάσεις, για συνθήκες, για κείμενα και όλα αυτά, αλλά υπάρχει και μια κουλτούρα, ένας λαός και μια παραδοσιακή διαχείριση που υπάρχει των πόρων. Και δεν είμαστε ικανοί να δεχτούμε ότι οι λαοί αυτοί υπάρχουν αλλά επειδή είναι σε κάποια μικρά νησιά δεν μας καταλαβαίνουν. Ο κόσμος αλλάζει. Και εμείς ενδιαφερόμαστε για την ανάπτυξη. Ο Λιβιέ, μήπως μπορείς να το δώσεις αυτό, να το περάσει από χέρι σε χέρι Κανείς δεν μιλάει για μια συνθήκη η οποία θα μας έδινε όχι ανταγωνιστικότητα, αλλά ένα πλαίσιο ζωής, μια ποιότητα ζωής, μέσω τέτοιου είδους αρωμάτων. Οι, άνθρωποι μας, οι λαοί μας, είναι πολύ ζωτικοί. Θέλουν να επιβιώσουν. Όχι μόνο σε σχέση με εσάς ή σε σχέση με ένα άλλο λαό, αλλά μόνο και μόνο μέσα στο περιβάλλον τους. Να σας δώσω και ένα άλλο προϊόν μας, για να σας δείξω ότι έχουμε προσαρμοστεί. Ε, είναι ε, λάδι από κοκοφίνικα, από καρίδα, λάδι καρίδας. Το PowerPoint που θα δείτε θα σας βοηθήσει απλώς να καταλάβετε καλύτερα αυτά που σας λέω. Και μετά επιστρέψτε μου παρακαλώ πολύ το στικ βανίλια που σα έδωσα. Ε, αν είσαστε και καλοί μαζί μου θα σας το αφήσω τελικά. Λοιπόν, προσπαθώ να σας αφυπνίσω ε, σε σχέση με το, με την ενοχελικότητα που επικρατούσε λίγο πριν, λίγο να κοιμηθούμε μερικοί από εμά. Αυτό το άρωμα της ε, βανίλιας, ε, του, της ε, καρύδας και αυτό το εθέριο έλαιο το οποίο έφερα επίση, α περάσουν από χέρι σε χέρι για να καταλάβετε ότι οι λαοί μα υπάρχουν, έχουν μία γλώσσα, έχουν μία παράδοση και δεν περιμένουν απλώς μία χιλιοστή, νιωστή καινούρια σύμβαση. Θέλουμε απλώς να ακούσετε την σιωπή που επικρατεί στους λαούς μας στον Ειρηνικό ωκεανό. Να σας ε, διαβάσω μερικές διαφάνειες. Το γεωγραφικό πλαίσιο της Πολυνησίας, ε, το συζητήσαμε προηγουμένως, ε, είναι πολύ εξαιρετική φύση γιατί είναι πολύ απομακρυσμένη η Πολυνησία. Υπάρχει μια ανάγκη ανανέωσης εταιρικής σχέσης. η ανανέωση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στους ανθρώπους και στον πολιτισμό τους, στο πλαίσιο μιας ε, παραδοσιακής διαχείρισης. Το ιεραρχικό πλαίσιο... Α, εδώ βλέπετε την Πολυνησία. Βλέπετε το βαθύ μπλε της Ευρώπης που ε, και η Πολυνησία πάνω από την Ευρώπη. Είμαστε πιο πολλοί αριθμοί από του Καλλιδόνιου, αντιθέτω από ό,τι είπε προηγουμένω. Αυτό είναι θέμα στατιστικό, όχι ε, εγωισμού. Ε, είμαστε πιο πολλοί αριθμοί από του Καλλιδόνιου. 10 ε, εκατομμύρια τρόνκα χιλιόμετρα, 5 εκατομμύρια ανήκουν στην Πολυνησία. 164 νησιά που κατοικούνται. Είμαστε ένας χώρος με εξαιρετική βιοπικιλότητα. Ε, το μικρό τραγουδάκι το οποίο σας έλεγα προηγουμένως υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός πάει χέρι-χέρι με τη βιοπικιλότητα. Μιλάμε ακριβώς για το ίδιο πράγμα. Δεν είναι φολκλόρ. Ε, στην Πολυνησία έχουμε τρεις διαφορετικές ώρες, ε, τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας. Ε, καταλαβαίνετε την έκταση ε, της περιοχής. Ε, γιατί χρειάζεται μια ανανέωση εταιρική σχέση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ευρωπαϊκό διαβατήριο, κάτι που μας επιτρέπει να μπαίνουμε και να βγαίνουμε ελεύθερα. Όχι όπω με τι ΗΠΑ. Γιατί η απικιακή ιστορία των χωρών μας μας χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα για εμπορικές σχέσεις Έχουμε ένα νόμισμα το οποίο συνδέεται με το ευρώ. Είμαστε οικονομικοί εταίροι και διαθέτουμε και, και εφαρμόζουμε και ένα μεγάλο τμήμα του οικονομικού κεκτημένου. Βέβαια η Πολυνησία έχει ε, δικές της αρμοδιότητες, ε, είναι αυτόνομη και με αυτή την έννοια ε, μπορούμε να διαλέγουμε το καλύτερο από ό,τι υπάρχει στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μας καινούργια σύνορα ή η συζήτηση είναι πολιτική και ιδεολογική, κοινωνική, ανθρώπινη, στην οποία ε, η κουλτούρα, ο πολιτισμός θα πρέπει να ξεπεράσει τα σύνορα. Νομίζω ότι αυτό το δεύτερο είναι καλύτερο. Τι ε, ταυτοποιεί αυτή τη στιγμή τη είχε. Είμαστε χώρες και εδάφη συνδεδεμένα, όπως σας είπα, με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι είχε σήμερα θα πρέπει να επεκταθούν, να μεγαλώσουν, ε, να διατηρήσουν μια πλέον ε, ε, μια σχέση ε, στενή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την εξελίξουν. Προτιμησιακή σχέση. Ε, γιατί μιλάμε ακριβώς. Πρόκειται για μια επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, σε, υπερπόντια, σε υπερπόντιες περιοχές Δηλαδή κατά βάση είναι μία ακόμα σύμβαση, μία ακόμα συμφωνία, κάτι που δύσκολα θα εξηγήσουμε στους πολίτες μας ότι είναι ενδιαφέρον και επικοδομητικό. Γιατί έτσι κι αλλιώς ε, νιώθουν ότι δεν καταλαβαίνουν όλες αυτές τις εξελίξεις. Ε, Παρ' όλα αυτά βέβαια, παρόλε τις δυσκολίες, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτε μας και να τους, ε, εξασφαλίσουμε συμμετοχή. Ε, ανταγωνιστικότητα. Αν η σύνδεση με τη ΣΥΧΕ ήταν μόνο οικονομική, τότε θα είχαμε πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Η δυνατότητα των πολυνήσεων, των ανθρώπων δηλαδή του ειρηνικού, με την ευρεία έννοια. Ε, να, σας έφερα τη βανίλια, το εθέριο έλαιο της βανίλιας, ε, το έλαιο κόπρα, όλα αυτά τα προϊόντα δείχνουν ότι υπάρχει οικονομικός δυναμισμός. Ε, προέρχονται αυτά τα δύο προϊόντα από την Μπόρα Μπόρα και από την Νησοτά. Βλέπετε ότι υπάρχει οικονομικός δυναμισμός, όμως αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Δεν περιμένουμε ότι κάποιο θα έρθει να μας φροντίσει. Όχι, δεν βρισκόμαστε σε τέτοιου κατάσταση. Υπάρχει και άλλο σύνδρομο εκτό τον οικονομικό. Έχουμε το απεικιοκό παρελθόν, έτσι, δύσκολο να επιληθεί, δύσκολο να ξεχαστεί, έχει αφήσει ίχνη, ανεξίτηλα. Ε, η ευρωπαϊκή αγορά είναι εξαιρετικά καλή για τέτοιου προϊόντα όπως τη βανίλια και το εθέριο άλωμα καρύδας, το κόπρα. Η προστιθέμενη αξία που μας δίνει η ευρωπαϊκή αγορά είναι τεράστια. Για μας είναι μεγάλη ευκαιρία. Είναι ευκαιρία η γυραιά Ήπειρος για την διακίνηση των προϊόντων μας. Έτσι ώστε η ανταλλαγή να μην είναι μονομερής μόνο, να είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν επιθυμούμε η Ευρώπη να είναι απλώς το ταμείο μας. Ούτε εμείς να είμαστε μόνο ζήτουλες χρημάτων. Η οικονομία έχει χρώμα. Για σας είναι πράσινη. Για μας είναι μπλε. Γαλάζια. Γιατί ζούμε από τη θάλασσα, μεγαλώσαμε στη θάλασσα, την τραγουδάμε. Μετακινούμαστε με πλωτά μέσα τα οποία ούτε μπορείτε να φανταστείτε εσείς εδώ μιλάμε για σκάφη που ε, διανύουν τεράστιες αποστάσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό ε, και τι σημαίνει μπλε οικονομία για μας, τι σημαίνει ψηλή τιμή του πετρελαίου κλπ. Χρειάζεται να μας γνωρίσουν. Για να ξεφύγουμε από αυτό το τυπο, αυτόν τον τυποποιημένο μύθο. Ο, ναι, ωραία πράσινα νερά, άσπρη άμμος ε, και μικρά νησιά μέσα του ωκεανού. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το πρότυπο και ε, σας έφερα αυτά τα προϊόντα εδώ πέρα για να σας δείξω ότι έχουμε και οικονομικές δυνατότητες να αναπτυχθούμε με διαφορετικό τρόπο. ένα προϊόν ξεπερνάει την οικονομική του διάσταση. Είναι και ένα από το, ενός πολιτισμού, μιας κουλτούρας. Θέλουμε όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και είμαι εδώ για να σας πείσω ότι υπάρχει κι άλλη μία εικόνα πέραν της ε, τυποποιημένης εικόνας τουριστικής που έχετε στο μυαλό σας. Άρα περιμένουμε από τις καινούριες συμβάσεις, από τα καινούργια κείμενα να το λάβουν υπόψη αυτό. Γιατί έχουμε βουνό από συμβάσεις και από κείμενα. Είναι πιο ψηλός ο πάκος με τις συνθήκες που υπάρχουν από το ύψος των υφάλων μας ε, που τριγυρίζουν τα νησιά μας γύρω-γύρω. Συνεπώ θα πρέπει οι καινούριες οι να χτιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και επειδή έχω γεράσει βάζω και γυαλιά, αντίθετα με τα όσα είπε η πρόεδρο, Βέβαια εξαιτία του υπολογιστή. Ε. Όπως πολλές χώρες, χαρακτηριζόμαστε και εμεί από μεγάλη βιοπικιλότητα. Ε, η εκμετάλλευσή τους όμως γίνεται πολύ συχνά από πολυεθνικές τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Μπορούμε να, βελτιώσουμε τους, να μειώσουμε τους κινδύνους. Ε, να... Οι επενδύσεις να γίνουν ε, επικοδομητικά στη χώρα μας. Μίλησα για τα γεωρικά προϊόντα, έχουμε τις υδατοκαλλιέργειες, ε, έχουμε βιοτεχνίες, οι πέρλες ας πούμε, τα τεχνητά μαργαριτάρια, είναι πολύ σημαντικό προϊόν και πάω ακόμα πιο γρήγορα, ε, είμαστε απομονωμένοι. Η απομόνωση αυτή, αντίθετα με τα όσα ενδεχομένω πιστεύει κανεί, δεν είναι μειονέκτημα. Ε, είναι πλούτος. Όταν κάποιο είναι απομονωμένο πάνω σε ένα νησί, καταλαβαίνει και κατανοεί καλύτερα, εκτιμά καλύτερα τον πλούτο τη βιοπικιλότητά του. Γιατί? Γιατί δεν είναι δυνατόν να πάει κανείς να κάνει ψώνια στο Καρφούρ ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο μεγάλο σούπερ μάρκετ. Οπότε χρειάζεται να αντλήσει ό,τι μπορεί από τη δική του παραδοσιακή κουλτούρα και να τη διαχειριστεί με έναν τρόπο βιώσιμο. Γι' αυτό το λόγο εξακολουθούμε να υπάρχουν. Εξακολουθούμε να υπάρχουμε. Είμαστε ε, ευάλωτοι. Το είπε η κυρία Γκρέσ προηγουμένως. Ενεργειακά για παράδειγμα. Ε, ε, η ε, πολεοδομία, αστιφιλία μας. Έχουμε πολύ αστιφιλία, οπότε δημιουργεί προβλήματα. Μεταφορές. Ε, ενέργεια λοιπόν, χωροταξία, μεταφορές. όλα αυτά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για μας. Ενεργειακά, για παράδειγμα, χρειάζεται να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας. Έχουμε θερμική ενέργεια, γεωθερμία. Βλέπετε εδώ το πελαμίς. Είναι ένα ε, προϊόν το οποίο μας ε, βοηθάει ε, να αναζητήσουμε το κρύο από τη θάλασσα το οποίο μόλις ε, ανεβεί στον, ε, στον αέρα δημιουργείται, δημιουργεί αέριο εξαιτία ε, του θερμικού σοκ με την επαφή με αέρα 26 βαθμών. Επίσης παράγουμε καύσιμα από φύκια για τις μεταφορές, την διαχείριση του νερού, των υδάτων που είναι απειλούμαστε από τις ε, πολυεθνικές αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά διαχείριση των υδάτων. Και ε, ω συμπέρασμα θα ήθελα να σας ε, ζητήσω συγγνώμη που ξεπέρασα κατά 3,5 λεπτά το χρόνο μου. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις, αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Παλαζή καταρχήν. Je je ne vous ai pas présenté M. Palazzi, mais M. Palazzi donc représente euh, une euh, très grande ONG. Ο κύριος Παλαζή εκπροσωπεί την Διεθνή Οργάνωση της Ευρώπης και μας εκπροσώπησε στα, στις νήσους ε, Ρεουνιών σε σχέση με θέματα βιοπικιλότητας. Euh, Καλημέρα σας και σας ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους διοργανωτές για την ακρόαση αυτή. Θα σας ε, υποβάλω επιπρόσθετα στοιχεία για το οικολογικό διακύβευμα των είχε. Όπως γνωρίζετε το 2008 στο Ρεουνιόν ε, διοργάνωσα την πρώτη διάσκεψη για τις είχε και τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες για θέματα βιοπικιλότητας. Ήταν ένα επίσημο θέμα της ε, υπογαλλική προεδρία. Τώρα εργάζομαι για μια, σε μια μεγάλη ΜΚΟ που έχει τη βάση της στις ΗΠΑ και στη Νέα Καλλιδονία. Αυτή η ΜΚΟ ασχολείται με, την, ε, με το διακύβευμα, τα οικολογικά διακυβεύματα στις ΙΧΕ. Βλέπετε εδώ στο χάρτη της ΙΧΕ υπάρχει μια παγκόσμια κατανομή, ανά δηλαδή, και πέρα από το διαφορετικό καθεστώς που της διέπει, βλέπετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο πολιτικών οντοτήτων που διασυνδέονται με την Ευρώπη. Επίσης υπάρχουν και τα καυτά σημεία της ε, βιοπικιλότητας, τα βλέπετε εδώ. Ε, υπάρχει μεγάλη επικάλυψη και η Ευρώπη συνδέεται με διάφορα σημεία βιοπικιλότητας. Όταν μιλάμε για σχέση καθαρού κέρδους, win-win, για τη βιοπικιλότητα, εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο ευεργέτημα για τους ε, αυτόχθονες μέσα στα πλαίσια αυτών των οικοσυστημάτων. Εδώ βλέπετε και τις χώρες ΑΚΕ στη Καραϊβική, στο Ειρηνικό, στον Ατλαντικό και βλέπετε τις δυνατότητες συνεργασίας, αυτά τα καυτά σημεία και συνεργασία που θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ είχε και χωρών ΑΚΕ. Ως προς ε, τις ειδικέ περιφέρειες, εδώ βλέπετε την Καραϊβική και έναν, ένα τρίτο των πολιτικών συστημάτων εντάσσονται στις ήχε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη απειλή στις, ως προς τις κλιματικές αλλαγές, γιατί δυστυχώς και οι κοραλιογενείς περιοχές έχουν υποβαθμιστεί και υπάρχουν πολλοί κυκλώνες και τυφώνες. Άρα οι χώρες της Καραϊβικής ε, διατρέχουν μεγάλους κινδύνους. Εδώ βλέπετε τον Ειρηνικό, βλέπετε τις ε, συστάδες νησιών στον Ειρηνικό, βλέπετε τις νήσους της Πολυνησίας, θα επανέλθω, τη Νέα Καλυδονία και εδώ βλέπετε τον πλούτο σε σχέση με την υπηρετική Ευρώπη ως προς τα είδη σε ψάρια βλέπετε ότι η Καλλιδονία έχει τα περισσότερα είδη σε σχέση με ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν επιδεινωθεί. Εδώ βλέπετε έμπρακτα πώς ισχύει αυτή η επιδείνωση. Υπάρχουν και ε, οι διάφορες υπηρεσίες των οικοσυστημάτων όπως η παροχή ύδατος, το πόσιμο νερό και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπετε τον Ινδικό, μιλάμε για τη Μαγιότ η οποία θα μετατραπεί σε πλέον απομακρυσμένη περιφέρεια. Και ως προς τη Μαγιότ θα ήθελα να σας πω ότι θα μετατραπεί σε πλέον απομακρυσμένη περιφέρεια και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την κατάσταση στη Μαγιότ, γιατί από είχε θα μετατραπεί σε πλέον απομακρυσμένη περιφέρεια, όπου θα ισχύσει μια ειδική ε, σύνδεση με, διαρθρωτικά, με τη συμμετοχή των ε, διαρθρωτικά, διαρθρωτικών ταμείων, Πρόκειται για μια ευάλωτη κατάσταση και η δημογραφική κατάσταση είναι εκρηκτική. Υπάρχει η μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού σε σχέση με ολόκληρο τον κόσμο και θα πρέπει να βελτιώσουμε την χρήση των υδάτων, ιδιαίτερα των υδάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να ανακυκλωθούν. Εδώ βλέπετε την ίσο Μαγιότ που επαπειλείται. Ως προς το νότιο Ατλαντικό βλέπετε ότι εκεί ε, ζουν Ευρωπαίοι κυρίως πολίτες και βεβαίως μίλησα και για την ε, περιοχή κάτω από την Αυστραλία. Βλέπετε την ίσο Άμστερνταμ εδώ και θα ήθελα να σας πω ότι χρησιμοποιείται αυτή η μέτρηση για τις, παγκοσμίως για τις ε, διάφορες μετρήσεις που γίνονται για τα αέρια τύπου θερμοκηπίου. Επί της νήσου Άμστερνταμ βρίσκεται αυτός ο σταθμός μέτρησης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ατού από επιστημονικής πλευράς για το μεσημβρινό ημισφαίριο. Εδώ βλέπετε τι γίνεται μέσα στο κτίριο, βλέπετε την οθόνη που κάνει τις μετρήσεις και έχουν γίνει πολλές μετρήσεις, βλέπετε τι κλιματικές έχουν, αλλαγές έχουν γίνει παγκοσμίω. Και εδώ η Γρυλανδία, που βλέπετε αυτό το τεράστιο κομμάτι, και καταλαβαίνετε ότι η Γαλλική Πολυνησία θα έχει μεγάλο πρόβλημα αν επέλθουν αλλαγές στη Γρυλανδία. Εάν δηλαδή βυθιστεί. Εδώ έχετε τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, τις υπερπόντιες και θα ήθελα να πω ότι έχουμε μεγάλες αλλιευτικές συμφωνίες. Εδώ βλέπετε τη Μαδαγασκάρη θα πρέπει να διαχειριστούμε τους ε, ωκεανούς. Εμείς ε, έχουμε τη δεύτερη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο την πέμπτη και βλέπετε το 20% των ωκεανών την χάνουν ευρωπαϊκής διαχείρισης. Σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα ήταν σκόπιμο να το δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί έχει μεγάλη σημασία για την παγκόσμια οικονομική διαχείριση των ωκεανών βλέπουμε ότι το 7% των κοραλιογενών περιοχών βρίσκονται στις ε, Ήχε. Μιλάμε για 300 εκατομμύρια ανθρώπων που βασίζονται στα κοράλια για την ε, καθημερινή τους επιβίωση. Όλα αυτά για να σας δείξω ότι το περιβάλλον έχει άμεση σύνδεση με τα υπερπόντια εδάφη. Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις. Εδώ βλέπετε το, την νήσο Ρεουνιών. Εδώ βλέπετε τις πυρκαγιές στη Νέα Καλυδονία, τις καταστροφές των ενδιατημάτων. Εδώ σας μίλησα για το περίφημο φυτό, το οποίο έχει εισβάλλει στο, στην ίσο αυτή και τα κοράλια έχουν μεγάλη σημασία και βλέπετε εδώ και τις νήσους και η Θα ήθελα να πάρω την Πολυνησία ως παράδειγμα, διότι έχει μεγάλη σημασία για τα οικοσυστήματα. Ας δούμε τα κοράλια. Μιλήσαμε για την παραγωγή βανίλιας και άλλες παραγωγές δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο, μεγάλος, ο μεγαλύτερος πυλώνας βασίζεται στις ε, κοραλιογενείς περιοχές. Εδώ βλέπετε θαυμάσια τοπία, μία θάλασσα τυρκουάζ, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από ένα ζωντανό οικοσύστημα που είναι τα κοράλια. Το ίδιο ισχύει και με τα σμαράγδια γιατί έχει μεγάλη σημασία για το εξαγωγικό εμπόριο. Ε, η αλία είναι βασική δραστηριότητα και από αυτήν εξαρτώνται πολλές ε, οικογένειες και εδώ έχουμε την, και την προστασία των παρακτήων περιοχών. Μιλάμε για επίπεδες νήσους, κατά κύριο λόγο, και βλέπετε ότι όταν έχουμε κοραλιογενείς υφάλους σε καλή κατάσταση μπορούμε να ζούμε ε, στο γυάλιο κύμα, στο θαλάσσιο κύμα. Αλλά αυτή η προστασία δεν υπάρχει όπου έχουν καταστραφεί οι κοραλιογενείς ύφαλοι. Και βλέπουμε εδώ ότι σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάμε για τρεις ατόλεις και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Πολυνησία διατρέχει μεγάλο κίνδυνο και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για τα αναπτυξιακά σχέδια στην Πολυνησία. Δηλαδή θα πρέπει να κρατήσουμε αυτά, αυτές τις ε, κοραλιογενείς, ε, τους κοραλιογενείς υφάλους. Όταν ε, η Γαλλία είχε την Προεδρία έκανε ορισμένες συστάσεις. Μιλήσαμε για την πρωτοβουλία BEST που ψήφισε το Κοινοβούλιο και μιλάμε για μία περίοδο δοκιμών, μία διετή περίοδο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την πρωτοβουλία BEST, γιατί τα υπερπόντια εδάφη σήμερα ε, δυστυχώς γνωρίζουν ένα μεγάλο κενό ως προς την χρηματοδότηση της βιοπικιλότητας δεν ξέρουμε πώς θα οριστεί η ειδική χρηματοδότηση, γιατί πολλές φορές λέμε ότι δεν μπορούμε να τους δώσουμε χρήματα από το Ταμείο Life, αλλά μπορούμε από το Ταμείο Best. Η βιοπικιλότητα όμως είναι μεγάλο διακύβευμα, είναι θέμα επιβίωσης αυτών των νήσων και θα πρέπει να την χάνουν ειδική χρηματοδότησης για να μπορέσουν να προστατεύσουν το οικοσύστημά τους. Το BEST ήταν ένα πολύ σημαντικό μέσο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, βοήθησαν στην δημιουργία του εδώ στην αίθουσα. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ γιατί πέρασα το χρόνο μου. Εδώ υπήρχε μία, έγινε μία έκθεση. Υπάρχει σε πολλές γλώσσες, είναι ένα κείμενο αναφοράς σε σχέση με τη βιοπικιλότητα και τις κλιματικές αλλαγές. Σε ένα λεπτό, ένα λεπτό, ούτε κανένα, θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να δούμε τα υπερπόντια διαμερίσματα μαζί με τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό θα πρέπει να το δούμε σε περιφερειακές συστάδες Επίσης, το περιβάλλον θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Μιλήσαμε για είδη τα οποία εισβάλλουν, για φυτά τα οποία εισβάλλουν σε συγκεκριμένες περιφέρειες και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Μιλάμε για χωροκατακτητικά φυτά, τα οποία βρίσκονται σε ορισμένες περιφέρειες και στην ουσία ακριβώς επειδή έχουν εισβάλλει το οικοσύστημα διατρέχει μεγάλο κίνδυνο και μιλάμε και για συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Ταμείο Life και εάν μπορούμε να βοηθήσουμε και με τη συμμετοχή του Life καθώς και του Best και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την εξέλιξη της νήσου Μαγιότ κατά τα ε, επερχόμενα έτη, διότι εδώ υπάρχει μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα και θα πρέπει να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Με συγχωρείτε που ξεπέρασα το χρόνο και σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να συζητήσουμε όλα, όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ε, δεν μπορούμε να... Ε, κάνουμε ερωταπαντήσεις ε, γιατί υπάρχει κι άλλος ένας ομιλητής 30 ε, δευτερόλεπτα θέλω μόνο θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής ποιες είναι οι συνέπειες ε, των πυρηνικών δοκιμών που θα μπορούσαν να είναι δραματικές κατά την άποψή μου για την βιοπικιλότητα και την κλιματική αλλαγή 30 δευτερόλεπτα μόνο παρακαλώ η απάντησή σας η κατάσταση δύο ατολών που χρησιμοποιήθηκαν για πυρηνικέ δοκιμές είναι εξή. Το κράτος αναγνωρίζει σήμερα τον κίνδυνο, αποδεδειγμένο κίνδυνο, ε, καταπώντησης ε, του ενός μεγάλου κομματιού μιας από αυτές τις ατόλες. Κάτι που κάτι που ε, προφανώς ε, ε, φορτώνει με ευθύνες τους ηθήνοντες. Αν τα νερά, αν το ύψος των νερών συνεχίσει να αυξάνεται με το σημερινό ρυθμό, θα τεθούν ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Στη Φουκουσίμα μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα ε, ψαρεύτηκαν τόνοι ανοιχτά της Καλιφόρνιας ε, με υψηλό ε, ραδιενέργεια, ραδιενέργειας, με υψηλό ποσοστό ραδιενέργειας. Συνεπώς καταλαβαίνετε ε, πώς η ραδιενέργεια μπορεί να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά σκεφτόμαστε αρκετά συχνά. Ευχαριστούμε. Περνάμε στο τρίτο πάνελ. Θα ζητήσω από τον κύριο Ντελατεριέ να πάρει το λόγο. Χαίρομαι που θα προεδρεύσω. Ε, καταλαβαίνετε καλύτερα νομίζω την προβληματική των είχε χάρη στις ε, παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων μέχρι τώρα. Στο πλαίσιο αυτού του πανέλ θα ανταλλάξουμε τις απόψεις, απόψεις για το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ΙΧΕ στην αντιξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές είχε είναι γειτονεύουν μάλλον με αναπτυσσόμενες χώρες, την Καρεβή και τον Ειρηνικό κυρίω, και θα μπορούσαν οι ΙΧΕ λοιπόν να αποτελέσουν λαμπαδιδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτές τις περιοχές. Ε, θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Ντελαντεριέρ που είναι πολιτικός ε, στη Νέα Καλλιδονία και φίλος. Είμαι σίγουρος ότι θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε έχετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μωρίς ε, Πόγκα που μου πρότεινε να κάνω μια παρουσίαση για αυτό το θέμα. Ασχολούμαι αυτό εδώ και πολλά χρόνια στη Νέα Καλλιδόνια. Δεν έχω το ταλέντο του κυρίου Μπριόν. Είμαι και τελευταίος στη σειρά, οπότε θα προσπαθήσω να μην σας ξαναρίξω σε υπνηλία. Να κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Είμαι υποχρεωμένος να ξανατονίσω ορισμένα πράγματα τα οποία έχουμε ήδη μιλήσει, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για περιφερειακή ολοκλήρωση αν δεν μιλήσουμε για οικονομική ανάπτυξη ή προστασία του περιβάλλοντος. Και δεν είναι περιττό ότι θα μας ε, επιτρέψει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Εγώ προέρχομαι από τον Ειρηνικό ωκεανό, από τη Νέα Καλλιδονία. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την Οκεανία, για εκείνη την περιοχή του κόσμου. Αλλά οι προτάσεις που κάνουμε εφαρμόζονται σε όλες τις ηχέ. Για να προετοιμάσω αυτή την παρουσίαση χρησιμοποίησα τα περισσότερα από τα ε, έγγραφα, ε, τα ε, ε, οποία, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Σαραμάντης ο κ. Σαραμάντης ε, και κάποια ε, έγγραφα της Γαλλικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Και βέβαια την πρόταση για τη νέα απόφαση σύνδεσης. Στα έγγραφα αυτά ο όρος που χρησιμοποιείται είναι ολοκλήρωση, περιφερειακή ολοκλήρωση. Το παράξενο βέβαια είναι ότι πουθενά σε κανένα από τα επίσημα έγγραφα δεν ορίζεται τι είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση. Θα μπορούσα να δώσω τον προσωπικό μου ορισμό βέβαια, αλλά θα προτιμήσω τη συμφωνία του, του, του Κοτονού, που έχει ένα ορισμό. Βέβαια αφορά πιο πολύ τις χώρες ΑΚΕ, αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη ΣΥΧΕ. Εκεί ο ορισμός είναι ο εξή. Ε, περιφερειακή ολοκλήρωση είναι η διαδικασία που ε, κάνει προσπάθεια να ε, ξεπεραστούν τα φυσικά, οικονομικά και προφαντικά προβλήματα των χωρών αυτών με συνεργασία στην χρήση των κοινών πόρων της περιφέρειας. Δηλαδή ε, είναι πιο ευρία από, πιο ευρύς αυτός ο ορεινός από τον ορισμό που δίδεται στις, ε, ε σχέσεις, ε, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης που περιορίζεται αυτός ο δεύτερος ορισμός στις ελεύθερες συναλλαγές. Όχι, η συμφωνία του Κοτονού περιέχει ένα ορισμό που λαμβάνει υπόψη παράγοντες πολύ σημαντικούς μέσω της ε, χρήσης του όρου ε, κοινά περιφερειακά αγαθά και κοινή περιφερειακή πόρη. Ε, όλα αυτά περιλαμβάνουν και τη βιοπικιλότητα, την εξαιρετική οικολογική, τον εξαιρετικό οικολογικό πλούτο των ΙΧΕ. Καταρχήν, ποια είναι τα τούτα πλεονεκτήματα των ΙΧΕ, μετά θα δώσω ένα απολογισμό της περιφερειακής ολοκλήρωσης και τρίτον, θα μιλήσω για την, ε, πώς πρακτικά θα μπορούσε να ενισχυθεί αυτή η περιφερειακή ολοκλήρωση. Ή είχε, έχουν ένα αριθμό από πλεονεκτήματα έτσι ώστε να είναι η ε, προφυλακή, εμπροστοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ε, ελέγχθη, οι ΙΧΕ έχουν ένα πόδι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα πόδι έξω αποτελούν τμήματα των ε, κρατών μελών, αλλά δεν αποτελούν τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Εξαιτία της, ε, το, το ότι ανήκουν σε ένα κράτο μέλος, όλοι οι κάτοικοι των ΙΧΕ είναι πολίτε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά στη Νέα Καλλιδονία έχουμε το προνόμιο να έχουμε τρεις ηθαγένειε. τη γαλλική, την ευρωπαϊκή και την καλλιδονιακή. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ε, παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι σε, όλες, σε όλα τα μέρη του κόσμου είχε και με αυτόν τον ε, τρόπο μπορούν ενώπιον όλων των τρίτων χωρών να προβάλλουν τις αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης και τις αρχές που είναι κοινέ για όλα τα κράτη-μέλη, θεσμικέ και άλλε αρχέ, ε, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, κράτο δικαίου και σεβασμός των, ανθρω... των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, οι ΙΧΕΕ έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες επίσης μπορούν να θεωρηθούν και πρέπει να είναι πλέον εκτίματα. Για παράδειγμα, ε, χαμηλή η μέση ηλικία του πληθυσμού, ε, υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης, πολιτιστικό πλούτο, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπριόν, πολύ ισχυρέ πολιτιστικέ ταυτότητε, αυτό αποτελεί πλεονέκτημα επίση. Έχουμε πόλου αριστεία ε, σε ορισμένα, σε ορισμένα, σε ορισμένα τομεί, ε, υποδομέ, ε, έρευνα, νοσοκομεία, τουρισμό κλπ. Όλα αυτά είναι κοινά χαρακτηριστικά αλλά το πιο κοινό είναι ο εξαιρετικός οικολογικός πλούτος η εξαιρετική βιοποικιλότητα Στη Νέα Καλλιδονία διαθέτουμε πάνω από 2.000 ενδυμικά φυτά και πάνω από 1.600 είδη ψαριών. Και τεράστιες υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές. Αν πάρουμε τις τέσσερις ηχέ του ειρηνικού Πολυνησία, ε, Wallis, Φορτούνα και Κέρν... καθώς επίσης και τη Νέα Καλλιδονία, παρόλο ότι αντιπροσωπεύουν το 6% του ε, πληθυσμού των 22 ε, ηχεία της περιοχής, καλύπτουν 30% της ε, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. σε, ε, στην βιοποικιλότητά τους ε, ε, είναι πραγματικά φυσικά εργαστήρια για να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Η διατήρηση αυτής της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι συλλογική υποχρέωση και η βιώσιμη εκμετάλλευσή τους αποτελεί, θα αποτελέσει οικονομικό πλεονέκτημα για το μέλλον. Παρόλα αυτά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα, ο απολογισμός ε, της ε, περιφερειακής ολοκλήρωσης, της, ε, της ολοκλήρωσης και ε, συμμετοχής ένταξης των ΙΧΕ εξακολουθεί να είναι πολύ φτωχός. Αυτό αναφερόταν και στην Πράσινη Βίβλο του 2008. Είναι σαφές ότι σε κανένα από τα έγγραφα που διαθέτουμε δεν βρίσκουμε λεπτομερή απολογισμό αυτής της περιφερειακής ολοκλήρωσης, περιφερειακή συνεργασίας. Ούτε καν σημαντικά παραδείγματα συγκεκριμένη υλοποίηση σε αυτό το τομέα. Η αξιολόγηση της ε, ε, περιφερειακής ολοκλήρωσης, της περιφερειακής συμμετοχής πραγματικά είναι κάτι για το μέλλον. Είναι κρεμότητα. Αν αναλύσουμε τα στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου, ιδιαίτερα στη στοιχεία τη Γαλλία, βλέπουμε ότι η εμπορικές ανταλλαγές με τις γειτονικέ χώρες είναι μικρές εξαιτία ενδεχομένως της ε, διαφοράς στο βιωτικό επίπεδο ε, και της διαφοράς στο οικονομικό επίπεδο, της επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Ε, επίσης διαπιστώνουμε ότι οι ανταλλαγές με τις Μητροπόλεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περισσότερες. Η Μητρόπολη είναι πάντοτε ο πρώτος οικονομικός και εμπορικός εταίρος ε, τον είχε. Η, η, είχε ε, συνδέονται με έναν τρόπο πολύ αδύναμο με τις χώρες ΑΚΕ, οικονομικά εννοώ. Ε, για τη Γαλλία, οι εξαγωγές προς την ε, προς τι χώρε ε, από τις ε, ηχέ τη Γαλλίας. Στι ΑΚΕ οι εξαγωγέ αποτελούν το 0,5% του ΑΕΠ του, ενώ οι εξαγωγέ το 2,2% του ΑΕΠ τους. Αντίθετα, οι ανταλλαγές με την Γαλλία, μεταξύ ηχέ της Γαλλίας και Γαλλίας, αντιπροσωπεύουν το 33% των συνολικών συναλλαγών. Βέβαια υπάρχει ένα διαφορετικό εμπορικό καθεστώς για τις ανταλλαγές με την Μητρόπολη από αυτό που υφίσταται για τις ανταλλαγές με τις χώρες ΑΚΕ. Ίσως αυτός είναι ένας λόγος. Πάντως χρειάζεται να ενισχυθούν οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις ΙΧΕ και τους γείτονές τους. Αυτός είναι ένας στόχος μακροπρόθεσμος βέβαια, αλλά θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να επιτευχθεί. Θα ήταν λανθασμένο να μην ακολουθηθεί ως προτεραιότητα. Τρίτο κομμάτι της παρουσίασής μου, υφίσταται μια συμφωνία, έτσι ώστε είχε να ε, γίνουν βιτρίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπροστοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά ε, είναι βέβαια προσευχές. Ε, ευχές και προσευχές θα πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Ε, πλέον. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από, το, από μια συγκεκριμένη οικονομική πραγματικότητα, από συγκεκριμένες αδυναμίες και πλεονεκτήματα, όπως αυτά που έχουμε εντοπίσει. Σε ό,τι αφορά την ε, περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων, ε, χρειάζεται να αναπτυχθούν οι εμπορικές σχέσεις, σαφέστατα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί και ευρωπαϊκά προγράμματα έτσι ώστε ε, να ενισχυθούν οι υποδομές μεταφορών και τηλεπικοινωνιών ε, καθώς επίσης και ενέργειας μέσω υποβρύχιων καλωδίων. Στο νότιο ειρηνικό διαπιστώνουμε ότι είναι πιο εύκολο να μεταβεί κανείς στην Ευρώπη, 18.000 μίλια μακριά, από ότι να πάει να παρακολουθήσει μία συνεδρίαση, ένα συνέδριο στην ίδια την Πολυνησία. Προτεραιότητα όμως θα πρέπει να δοθεί στην διαχείριση και διατήρηση ε, κοινών αγαθών και κοινών πόρων. Μιλώ για τη βιοπικιλότητα, το κλίμα, την, δια, την διαχείριση αποβλήτων, τις, ε, ε βιώσ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την προστασία των κορολογιωνών υφάλων, ε, ή την προστασία έναντι των φυσικών καταστροφών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις προτάσεις της Κομισιόν ως άξονας προτεραιότητας. Στην πράξη αυτό θα σήμαινε ενδεχομένως την δημιουργία κέντρων ε, αριστείας στις ΙΧΕ έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία στην έρευνα και την διατήρηση. Σε ό,τι τον τομέα της αλίας. Με τους φίλους από την Πολυνησία είδαμε τη σημασία αυτού του τομέα και είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε μέτρα, μέσα, κοινά μέσα ε, ε, επιτήρησης των θαλασσών και ε, αντίθετα ό,τι κάνουμε με το Βανουάτου που είναι χωρακέ, ε, ε, μάλλον όπως κάνουμε με το Βανουάτου ε, που έχουμε κοινά μέσα για την ε, ε, για την παρακολούθηση των θαλασσών. Επίσης, έχουμε ζήτημα ε, κυκλώνων και γενικώ καιρικών φαινομένων, τα οποία πλήττουν όλη την, όλες περιοχές. Έχουμε μέχρι και κλιματικούς μετανάστες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα λογισμικό για την συνεργασία, περιφερειακή συνεργασία σε αυτά τα θέματα θέματα περιβάλλοντος. Το 2009 δημιουργήθηκε η, η, πλατφόρμα για διαχείριση κινδύνων, περιβαλλοντικών καταστροφών στην Οκεανία και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ο χρόνος με πιέζει. Θα μπορούσα επίσης να αναφέρω την, ε, ε, την επιχείρηση ε, ανάπλασης κατόπιν ε, φυσικών καταστροφών ε, έχουμε Φίτζι και Βανουάτου, δύο χωρίς και δύο, χωρίς, και δύο ΙΧΕ, Πολυνησία και Νέα Καλλιδονία, ε, που συνεργάστηκαν για την ανάπλαση των φυσικών και ανάκτηση των φυσικών πόρων μετά από φυσικές καταστροφές. Επίσης, ένα πρόγραμμα περιφερειακής συνεργασίας για την διατήρηση των παραθαλάσσιων περιοχών, παραθαλάσσιων νησιωτικών περιοχών. Ε, επικεφαλής ήταν η Πολυνησία, είναι ένα πρόγραμμα ε, ε, που ονομάζεται Integr. Είναι ένα πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Αναπτυσιακό Ταμείο, 12 εκατομμύρια ευρώ, τέσσερα ησυχία από το Νότιο Ειρηνικό, Πολυνησία, ε, Πολυνσία και Νέα Καλυδονία συμμετέχουν. Ε, αυτές οι τέσσερις ΙΧΕ θα συνεργαστούν με την Επιτροπή του Ειρηνικού, που είναι μια περιφερειακή οργάνωση, και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Integra, λοιπόν. Αυτό το σχέδιο έχει ως στόχο να ενισχύσει την ολοκληρωμένη διαχείριση ε, των ε, παραθαλάσσιων νησιωτικών περιοχών ε, σε ηχέ του Νότιου Ειρηνικού. Είναι απαραίτητο λοιπόν στην μελλοντική απόφαση σύνδεσης να καθοριστεί μια πραγματική στρατηγική, κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στρατηγική περιφερειακής ε, ολοκλήρωσης και γι' αυτό το λόγο τα περιφερειακά και τα εδαφικά ε, προγράμματα θα πρέπει να είναι το εργαλείο αυτής της στρατηγικής. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ε, το, την πρόταση του Γαλλικού Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου να δημιουργηθεί ένα ταμείο που θα χρηματοδοτεί τρίτες χώρες με ποσά παρόμοια με αυτά που χρηματοδοτούνται ΧΕ έτσι ώστε οι τρίτες χώρες να μπορέσουν να συγχρηματοδοτήσουν κοινά σχέδια με τις πλέον περιφερειακές περιοχές Ευρωπαϊκής ΕΕ και με τις ΧΕ. Είναι μία από τις προτάσεις για την, που υπάρχουν για την περιφερειακή χρηματοδότηση και θα ήθελα να τη λάβει υπόψη η Κομισιόν. Οι ΙΧΕ έχουν κοινέ αρχές και, και κοινέ αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει πάνω στη ΙΧΕ μια πραγματική πολιτική ευρεία γειτονία, ε, που θα βασίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ε, μιλάμε πιο πολύ για αξίες και κανόνες παρά για χρήμα. Συνεπώς μέσω των ΙΧΕ θα πρέπει να προωθηθούν και να διαφημιστούν οι αρχές και οι αξίες και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει τα συμφέροντα των ΙΧΕ να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη στις συμφωνίες και συζητήσεις που γίνονται διμερός και πολυμερός με τρίτες χώρες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Ε, θα πρέπει να ε, συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες και γιατί να μην κάνουμε αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη με τις ΙΧΕ τους. Δηλαδή να τους εκχωρήσουμε αρμοδιότητες έτσι ώστε οι ίδιοι εκπρόσωποι των ΙΧΕ να είναι διαπραγματευτές. Τέλος, να πω ότι η μελλοντική απόφαση σύνδεσης θα πρέπει να ξεκινήσει μια στρατηγική ε, περιφερειακή ολοκλήρωση που θα βασίζεται σε δύο άξονες. Πρώτον, εταιρική σχέση και δεύτερον, συνευθύνη, συνυπευθυνότητα. Ανάμεσα στι ΙΧΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας, κύριε Ντελαντριέρ. Δεν έχουμε πια χρόνο για υποβολή ερωτήσεων. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκρές για να συνοψίσει. Κύριε Πόγκα, δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρεμβαίνοντες και όσους, όλους όσους προσήλθαν. Λυπάμαι που δεν ήμασταν περισσότεροι, αλλά νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων ήταν ε, άκρος χρήσιμη και θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη καλύτερα ε, όλες αυτές τις διαστάσεις που ε, αναφέρθηκαν εδώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.